Ε, ε, Καλώς ορίσατε κυρία Τάισον, υποψήφια επίτροπος για απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δεξιότητες και κινητικότητα του εργατικού δυναμικού η επιστολή του υποψηφίου Προέδρου του κ. Ζαν Κλοντ Γιονκέρ του είπε ότι θα συμβάλει η κυρία Τάισον να εφαρμόσει συντονισμένα προγράμματα, αυτά που συντονίζονται τον Αντιπρόεδρο για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας και τον Αντιπρόεδρο για την Ευρώπη και τον κοινωνικό διάλογο. Θα συνεργάζεται στενά με τον Επίτροπο Οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων, φορολογήσης και τελωνίων. Η κυρία Τάισεν θα έχει υπηρεσίες υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Συμπερίληψη, Ένταξη. Θα την βοηθήσουν όμως και οι κάτω μονάδες μεταρρυθμίσεως της αγοράς εργασίας, δεξιοτήτων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης και πολιτικής για την εκπαίδευση των ανηλίκων και δικαιώματων ατόμων με, ειδικές, με αναπηρίες, καθώς και θα επικουρείται και από τη Eurostat. Θα είναι υπεύθυνη και για σχέσεις με τέσσερις υπηρεσίες αρμόδιες για τον τομέα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και την υγεία, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη πρόθεση επαγγελματική κατάρτιση στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωση και εργασία και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτιση. Σύμφωνα με τι κατευθυντήριε γραμμέ για την έγκριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους υποψήφιους επιτρόπους επί τη βάση και παραθέτω γενικών ικανοτήτων αφοσίωση τον ευρωπαϊκό σκοπό και προσωπική ανεξαρτησία. Θα αξιολογήσει τη γνώση των μελλοντικών τους χαρτοφυλακίων και των διαφόρων ικανοτήτων τους όσον αφορά την επικοινωνία. Πριν την ακρόση, να πω ότι έχετε απαντήσει γραπτός, κυρία Τάισον, στα προπαρασκευαστικά ερωτηματολόγια οι γραπτές απαντήσεις έχουν διανεμηθεί στα μέλη σε όλες τις γλώσσες οπότε είμαστε όλοι καλά προετοιμασμένοι για τις ερωτήσεις που θα σας θέσουμε προφορικά. Κάποια λόγια για την, την όλη δομή της ε, συζητήσεως η κυρία Τάισον καλείται να κάνει μια εναρκτήρια προφορική δήλωση. Δεν θα είναι μεγαλύτερη από 15 λεπτά. Θα έχει 5 λεπτά στο τέλος της συνεδριάσεως για να ολοκληρώσει την παρουσίασή της. Μετά αυτή την εισαγωγή θα υποβληθούν 45 ερωτήσεις από ευρωβουλευτές. Η συζήτηση θα διεξαχθεί σύμφωνα με την διαδικασία ping-pong όπως αποκαλείται ε, ο καθένα θα έχει τρία λεπτά στη διάθεσή του. Μάλλον, ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση. Τρία λεπτό για την ερωταπάντηση. Έχουμε μεγάλο αριθμό ερωτήσεων και γι' αυτό πρέπει να σεβαστείτε σας παρακαλώ ε, με αυστηρότητα το χρονικό όριο. Θα, θα επιβάλλω τον κανόνα. Αν ο μιλητής απουσιάζει, στο χρόνο που προβλέπεται ότι τεθεί, δεν θα υποβληθεί το ερώτημά του, δεν θα υπάρχει διαδικασία catch the eye. Και η Επιτροπή Απασχόλησης είναι η καθήλια αρμόδια επιτροπή για την ακρόαση. Αλλά έχουμε και την Επιτροπή Πολιτισμού και την Επιτροπή Γυναικών που θα συμμετάσχουν στην ακρόαση ε, που ασχολούνται, καλύπτουν και αυτές το θέμα. Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους και από αυτές τις δύο επιτροπές και όπως αναφέρεται στον κατάλογο των αγορητών θα θέσουν διάφορες ερωτήσεις που σχετίζονται με τις εντολές και τις αρμοδιότητες των επιτροπών. Ο πρώτος γύρος ερωτήσεων ανήκει στους συντονιστές και έναν εκπρόσωπο των μη εγγραμμένων μελών. Η διερμηνία ε, παρέχεται σε 23 γλώσσες. Όλοι οι ομιλητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα τους το ίδιο θα κάνω και εγώ σύντομα. Να υπενθυμίσουμε στους ομιλητές ότι αυτό που θα πούν πρέπει να μεταφραστεί μέσω των διερμηνέων. Άρα θα ήταν καλό να μην μιλάμε πολύ γρήγορα. Η κυρία Τάισεν ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει την μητρική της γλώσσα, τα Ολλανδικά, για τις απαντήσεις το επιχείρημά της είναι ότι θέλει να είναι όσο πιο ακριβής γίνεται και σαφής. Οι παλαιότεροι συνάδελφοι γνωρίζουν την κυρία Τάισεν κατέχει ε, πλήρως και την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. Θα μεταδίδεται στο διαδίκτυο ζωντανά στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η συνεδρίαση και θα μπορείτε να βλέπετε και μαγνητοσκοπήσεις ε, της ακροάσεως στην ίδια ιστοσελίδα. Θα μιλήσω τώρα τη μητρική μου γλώσσα, σου ειδικά. Θα σας δώσω, θα προβώ σε κάποια αρχικά σχόλια προσωπικής ε, φύσεως που αφορούν την ακρόαση. Ένας, μία από τις ε, πιο έντονες αναμνήσεις από τις εκλογές, ευρωεκλογές φέτο ήταν ένα τηλεφώνημα που έλαβα από έναν ιερέα που εργάζεται για την Σουηδική Εκκλησία, μία ιερέα, στη Νότια ε, Σουηδία, ανησυχούσε πολύ ιερεύς και ήταν απελπισμένη για τη φτώχεια που είδε ε, σε ένα χώρο στάθμευσης ε, στην πόλη της. Έβλεπε σειρά φορτηγών που περίμεναν νέες παραδόσεις και καμιά φορά οι οδηγοί των φορτηγών ζούσαν και ζουν στα φορτηγά, κανείς δεν είχε συλλογική σύμβαση ή ε, κάποια προστασία, δεν πληρωνόταν όταν δεν οδηγούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαν να πάνε στο σπίτι τους όμως. Περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα όσον αφορά την υγιεινή και τα τρόφιμα και όπως ξέρετε ο χειμώνα μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληρός στη Σουηδία. Κάποιοι από αυτούς έπρεπε να προστατευθούν έχοντας ε, μικρές ε, θερμάς, μικρές σόμπες κατασκήνωσης. Ήταν πολύ δύσκολο να κρατάνε τις μηχανές αναμένες για να ζεσταίνονται. Αυτή είναι η κατάσταση στον τομέα των μεταφορών και σε πολλούς άλλους τομείς στην Ευρώπη. Είναι κάτι που το βλέπουμε και με γυναίκες εργαζόμενες σε πολλούς τομείς. Αυτή είναι η κατάσταση, η σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη όπου τα δικαιώματα των ανθρώπων και όλοι οι κανόνες έχουν ε, θρηματιστεί λόγω της κρίσης. Και εκείνοι που θέλουν να εργαστούν δεν είναι απλώς άνεργοι, δεν έχουν καν δικαιώματα. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πόρα απέχει από τους στόχους της για το 2020. Πάνω από 120 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν με φτώχεια κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρώπη. 32,4 εκατομμύρια είναι παιδιά. Ε, τον Ιούλιο φέτος η ανεργία των νέων ήταν στα 22% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλές διακυμάνσεις μεταξύ κρατών μελών. Σε κάποιες χώρες είναι τόσο ψηλό το ποσοστό που πάνω από το μισό των νέων της χώρας ε, είναι άνεργοι. Και είδαμε τις συνέπειες αυτού. Το είδαμε και στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών φέτος. Το βλέπουμε όταν βλέπουμε ποιος είναι ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης ε, εκφράζεται η απογοήτευση, η απελπισία και απευθύνονται προς αντιδημοκρατικά κόμματα και ακρεφνή κόμματα ε, οι άνθρωποι. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει το 2014 στην Ευρώπη. Σκοπός μας την επόμενη πενταετία είναι να λύσουμε τα προβλήματα της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη και να δημιουργήσουμε νέες βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. Δεν θέλουμε να υπάρχει ανταγωνισμό σε χαμηλές αμοιβέ και κακές συνθήκες. Ε, θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, να λύσουμε τα προβλήματα. Ο καθένας να έχει τις ίδιες δυνατότητες και να έχουμε ισχυρή αγορά εργασίας. Άρα ε, πρέπει να, πρέπει να κινηθούμε στεναρά. Και ο νέος επίτροπος του τομέα έχει πάρα πολλές ευθύνες για τον χώρο αυτό. Εγώ προσωπικά και οι άλλοι πολίτες της Ευρώπης περιμένουμε η κυρία Τάισεν αρκετά σκληρή και ευφυής, ούτως ώστε να ε, εκτελέσει αυτά τα πολύ σημαντικά καθήκοντα, να είναι αρκετά δυνατή, ούτως ώστε να επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές. Είναι, δεν είναι πια η ώρα να καθόμαστε να περιμένουμε, είναι ώρα για δράση τώρα. Σε αυτή τη φάση θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Τάισεν να κάνει μια εισαγωγική παρέμβαση, να δούμε ποιες φιλοδοξίες έχει και ποιε δράσεις θέλει να δρομολογήσει. καλώ ήρθατε για μια ακόμη φορά και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Okay. Excuse me. Honorable Chair τιμή, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Στη ζωή είναι σημαντικό να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, χωρίς ε, επεκφυγές. Σήμερα, 26 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χωρίς θέση εργασία. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό. 7,5 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι μεταξύ 15 και 24 δεν είναι ούτε σε κάποια θέση απασχόλησης, ούτε σε κάποια θέση εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε και πάνω από 124 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με την φτώχεια ή με την κοινωνικό αποκλεισμό. Ούτε αυτό μπορούμε να το αποδεχτούμε. Γι' αυτό λοιπόν η στόχη μου για τα επόμενα πέντε χρόνια είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Να αγωνιστούμε για πιο πολλές θέσεις εργασίας, για καλύτερη κοινωνική προστασία, και να καταπολεμήσουμε την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτές είναι οι προτεραιότητες πολλών Ευρωπαίων και είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι αυτές είναι και οι δικές σας προτεραιότητες. Αγαπητοί συνάδελφοι, ως μέλος του Κοινοβουλίου αυτού για 23 περίπου χρόνια, ο σεβασμός μου για το θεσμικό αυτό όργανο έχει αυξηθεί διαρκώς και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανεί τη δέσμευσή μου για μια καλύτερη Ευρώπη. Εδώ, στο Κοινοβούλιο, με λόγια αλλά και πράξεις, πάντα ήθελα να υποστηρίξω την προόδο της Ευρώπης με συγκεκριμένα αποτελέσματα όμως για τον άνθρωπο. Και αυτό πάντα το έκανα βάσει ε, πλειοψηφιών, με ευρεία υποστήριξη. Και θα ήθελα να υποδείξω ότι οι δύο τελευταίες μου εκθέσεις σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Υποπτία και την μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αλλά και η δεσμευσή μου την εποχή εκείνη για να βρω μια πλειοψηφία για αυτή την οδηγία αλλά και για να υπάρξει κοινωνικός προσανατολισμός. Πάντα λοιπόν ε, λειτουργούσα πέρα από τα όρια των συνόρων, των εθνικών συνόρων, των ομάδων και πάντα σε πιστή συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα. Και αν με τη δική σας έγκριση διοριστώ ως Επίτροπος για τις απασχόλησης και κοινωνικές υποθέσεις ε, και κινητικότητα, σίγουρα θα συνεχίσω να απευθύνομαι σε αυτές τις ε, προκλήσεις. Η χρηματοπιστωτική κρίση είχε σκληρό τίμημα και τα έκτακτα μέτρα τα οποία αναγκάστηκε να πάρει η Ένωση για να καταπολεμήσει την κρίση ήταν απαραίτητα. Τώρα διαφέρονται σιγά σιγά οι θετικέ επιδράσεις ε, της πολιτικής αυτής, σιγά σιγά και αντιστακτικά. Αλλά την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων, είναι, αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε μπορέσει ακόμα να το πετύχουμε. Γι' αυτό λοιπόν η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πετύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θα έχουν απτές συνέπειες για όλους τους πολίτες. Ο πρόεδρος Σαν Γιούνκερ μου ζήτησε να φροντίσω προκειμένου η λέξη κοινωνικός να ξαναποκτήσει την πλήρη σημασία της και να ολοκληρωθεί η οικονομία της αγοράς πλήρως. Α, αυτή την πρόκληση την αποδέχομαι γιατί είμαι πεπισμένη υποστηρίκτρια της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς όπου η ελευθερία, η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη ε, συνυπάρχουν. Είναι λοιπόν σαφές ότι θα πρέπει να είναι ο στόχος μας η επόμενη επιτροπή θα πρέπει και σε κοινωνικό επίπεδο να έχει απτά αποτελέσματα από το ο κοινωνικής απασχόλησης απασχόλησης κοινωνικών υποθέσεων, ικανοτήτων και εργασιακής κινητικότητας. Θέλω λοιπόν να φροντίσω να το πετύχουμε αυτό μαζί με τους ε, υποψήφιους ε, αντιπροέδρους και επιτρόπους, ιδιαίτερως με τους συναδέλφους Κατάριν Νομπροβόσκης και Μοσκοβίτση, θα δουλέψουμε ως μία ομάδα και θεωρώ ότι θα είναι δική μου, δικό μου καθήκον προκειμένου να φροντίσουμε τα επόμενα πέντε χρόνια η πολιτική σε όλους τους τομείς να λάβει υπόψη όλες τις κοινωνικές επιπτώσεις των μέτρων. Όπως ε, είπε ήδη ο Jean-Claude Juncker, δεν θα έχουμε εξέλθει από την κρίση όσο 26 εκατομμύρια συμπολιτών μας εξακολουθούν να παραμένουν άνεργοι. Κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή μεταξύ ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής ισότητας. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος που από κοινού αποτελούν το βάθρο της ε, κοινωνικής οικονομίας της αγοράς που είναι ανταγωνιστική και αλληλέγγυα. Ο ρόλος μου θα είναι να συμβάλλω στη διαμόρφωση των καλύτερων προϋποθέσεων για να επιστρέψουν οι άνεργοι στην αγορά εργασίας και να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και την φτώχεια. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας αγοράς εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας αγοράς εργασίας που θα είναι δυναμική και ολοκληρωμένη εκεί που οι ετούντες θέση απασχόλησης θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επιχειρήσεων όπου και αν βρίσκονται αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία κατάρτιση που θα πρέπει να είναι προσιτή σε όλους, να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες, να επικεντρώνεται ιδιαίτερα στους μακροχρόνια άνεργους και στην κινητικότητα των εργαζομένων. Όλα αυτά είναι απαραίτητα μέτρα σήμερα για την Ευρώπη για να ξαναβρούμε το δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης και να μειώσουμε τη φτώχεια. Όσες και όσοι με γνωρίζουν, γνωρίζουν κάλλιστα ότι δεν ψάχνω ποτέ απλοϊκές λύσεις για περίπλοκα προβλήματα. Κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε αξιόπιστο, ούτε έντιμο, αλλά ούτε και αποτελεσματικό. Θέλω απτά αποτελέσματα. Θέλω οι επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να προσαρμόζονται στις ραγδαίες εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης, στην οποία συμμετέχουμε ενεργά. Θέλω ταυτόχρονα εργαζόμενοι και εργοδότες να συμβάλλουν με την εργασία τους στην δημιουργία πλούτου, με προϋποθέσεις όμως που θα εξασφαλίζουν την αξιοπρέπειά τους τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και την ισότητα των ευκαιριών. Άνδρες και γυναίκες, υπήκοοι της χώρας στην οποία απασχολούνται ή άλλης χώρας, ανάπηροι, όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και όλοι έχουν δικαίωμα και αξίζουν ίση αμοιβή για ίσες υπηρεσίες για ίση εργασία. Εξάλλου, η διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητάς μας και η διαχρονικότητα των κοινωνικών συστημάτων προστασίας μας απαιτούν την, τον εντοπισμό των καταχρήσεων και την ε, τιμωρία τους. Γι' αυτό θα ε, δώσω έμφαση σε τέσσερις προτεραιότητες που έχουν ίση σημασία και αυτές θα προσπίσω. Καταρχήν, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πολλές θέσεις εργασίας ε, έχουν καταστραφεί, καταρακωθεί από την κρίση. Εκατομμύρια. Για να δώσουμε λοιπόν νέες προοπτικές στους ανέργους, θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται ευνοϊκές ε, συνθήκες για να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, είτε παραδοσιακές είτε καινοτόμες, και να κατακτήσουν νέες αγορές. Δεύτερον, πρόσβαση στην απασχόληση. Μία μαζική απασχόληση συνυπάρχει με ένα γεράσκον εργατικό δυναμικό και, και με ανέργους, κυρίως νέους, που συχνά είναι ανειδίκευτοι, δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και δεν έχουν πια πρόσβαση σε σταθερές ε, θέσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν περαιτέρω προσπάθειες για να καθοδηγήσουμε και να προσανατολίσουμε τους νέους και να επιτρέψουμε στις γυναίκες και στους αναπήρους πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Και επίσης να επανενεργοποιήσουμε τους μακροχρόνια άνεργους. Μεταξύ των λύσεων που προτείνω είναι μια καλύτερη κινητικότητα των εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν αυτή την κινητικότητα να την προωθήσουμε. Τρίτον, δεξιότητες, προσόντα. Η ανταγωνιστικότητά μας εξαρτάται πρώτα απ' όλα από τις δεξιότητές μας. Οι εργαζόμενοι σήμερα στη διάρκεια του ενεργού τους βίου έχουν πολλές επαγγελματικές σταδιοδρομίες. Θέλουμε λοιπόν να καλύψουμε τις καθυστερήσεις τους και τα κενά τους στην απόκτηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσόντων ε, για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους ασχέτως της ηλικία τους. Τέταρτον, η κοινωνική προστασία. Η κοινωνική προστασία είναι θεμελιώδης επένδυση και βάση της ευημερία μας. Το 2010 διατυπώσαμε ένα ξεκάθαρο στόχο, ότι μέχρι το 2020 θέλουμε να μειώσουμε κατά 20 εκατομμύρια τον αριθμό των ανθρώπων που είναι θύματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Δυστυχώς το αντίθετο συνέβη. Η κρίση οδήγησε σε μια απότομη αύξηση της φτώχειας και του αποκλεισμού τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας που έχουμε θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά και καλύτερα προσανατολισμένα στα αποτελέσματα, διασφαλίζοντας μια εφορία μακροπρόθεσμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, για να υλοποιήσουμε τις προτεραιότητες αυτές θα χρησιμοποιήσω όλα τα μέτρα και τους μηχανισμούς που έχω στη διάθεσή μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα επικεντρωθώ κυρίως σε τέσσερις άξονες. Πρώτον, Κινητοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων. Στόχος μου είναι να προωθήσω τις επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να βοηθήσω στην επαναφορά των ανέργων στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό και θα συνεργαστώ με τον Αντιπρόεδρο Γύρ και Κατάινεν για να ετοιμάσουμε την κινητοποίηση 300 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύσεων που έχει αναγγείλει ο Ζανκλώδ Γιουνκέρ. Σας διαβεβαιώ ότι θα κινητοποιήσω όλα τα διαθέσιμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία και μηχανισμούς για να επενδύσουν στους ανθρώπους. Ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Ενίσχυσης στους Απόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Όλα αυτά τα ταμεία και τα κονδύλια τους θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, δημιουργία δεξιοτήτων και καταπολέμηση τη φτώχεια. Επίση, θα επιταχύνω την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε σάρκα και οστά στο, στα προγράμματα για την εγγύηση για την νεολαία. Δεύτερον, η οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει ταχύτητα. Η απασχόληση και οι κοινωνικέ πολιτικέ θα πρέπει να είναι πιο παρούσε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα συνεργαστώ λοιπόν στενά με τον Αντιπρόεδρο Βάλτη Ντομπρόφσκη και τον συνάδελφο Μοσκοβισή ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνουμε να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η ευάθυνση των μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη είναι απαραίτητη. Αλλά κάτι τέτοιο προϋποθέτει μεγαλύτερη δικαιοσύνη και βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων. Ο κοινωνικός αντίκτυπος ε, των ε, προγραμμάτων διάσωση για εύθευστε χώρε θα πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό το στόχο. Επίση, θα πρέπει να επανακινήσουμε τον κοινωνικό διάλογο. Θα συνεργαστώ με τον Αντιπρόεδρο των ώστε οι εργαζόμενοι και οι εργοδότε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνουν πραγματικοί εταίροι μα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Οι σημαντικέ και δύσκολε κοινωνικέ μεταρρυθμίσει θα πρέπει να συζητηθούν πλήρω με του κοινωνικού εταίρου και να εμπλέκουν όλους τους βασικούς φορείς ε, και να καλύπτουν όλο το οικονομικό και κοινωνικό φάσμα συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη σήμερα. Τρίτον, αναλογικότητα στους κοινού κανόνες. Έτσι θα δημιουργήσουμε συνθήκες ίσου ανταγωνισμού και θα προσπίσουμε την ενιαία αγορά χωρίς να δημιουργούμε υπερβολικό άχθος για τους διάφορους φορείς. Θα συνεργαστώ στενά με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσω μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτό το σημείο θα πρέπει να ενισχυθεί. Και σύμφωνα με, την, με το πρόγραμμα για την έξυπνη νομοθεσία, θα αξιολογήσω την υφιστάμενη νομοθεσία προκειμένου να είναι αποτελεσματική, αναλογική και εύχρηστη, εύκολης εφαρμογής. Θα πρέπει επίσης να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους από νέους κινδύνους και γι' αυτό θα προτείνω τον εξυγχρονισμό και όπου δει και την απλούστευση του νομοθετικού μας κεκτημένου, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίσω ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Θα εξετάσω και θα υποβάλω και νέες πρωτοβουλίες όπου χρειάζεται, για παράδειγμα στο θέμα της κινητικότητας των εργαζομένων. Τέλος, καθήκον μου είναι να αξιοποιήσω στο έπακρο τους μηχανισμούς και τις εταιρικές σχέσεις που έχουμε και τα επόμενα χρόνια από κοινού και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη, με τους κοινωνικούς εταίρους και τους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη πιο δίκαιη και πιο βιώσιμη. Την επόμενη πενταετία θα έχω στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα είμαι στη διάθεσή σας για να συζητούμε τακτικά την πορεία των εργασιών μας. Έχουμε ένα κοινό στόχο. Τους ανθρώπους, την υγεία τους, την δουλειά τους, την ευμάρειά τους. Η Ευρώπη είναι για τους ανθρώπους και μπορείτε να υπολογίζετε σε μένα. Θα είμαι ο σύμμαχός σας για να πραγματώσουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πολύ κυρία Τάισεν. Θα δώσω το λόγο τώρα στα μέλη σύμφωνα με τον κατάλογο των ομιλητών. Άρα δίνω το λόγο στον κύριο David Κάζα του ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υποψήφια Επίτροπε, στην εισαγωγική σας ομιλία τονίσατε επανειλημμένα και σωστά, πιστεύω, ότι η δημιουργία θέσεις απασχόλησης, θέσεων απασχόλησης πρέπει να είναι προτεραιότητα. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι ανέργοι, εκατομμύρια νέοι. Κάτι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε. Η υποστήριξη των ανέργων και στήριξή τους να βρουν δουλειά είναι πολύ σημαντικό θέμα. Στο χαρτοφυλάκι όσα αντιθέτεται πολλά μέσα που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση αντιμετώπιση του προβλήματος δεξιοτήτων με θέσεις εργασίας, να μην ταιριάζουν, να κινητοποιηθούν τα διάφορα δημοσιονομικά εργαλεία, όλα αυτά είναι καλά. Αλλά εκείνοι που είναι πρόθυμοι να εργαστούν, δεν, οι βούληση να δεν αρκεί. Πρέπει να είναι διαθέσιμες οι θέσεις απασχόλησης. Τι σχεδιάζει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δημιουργήσει σωστές περιστάσεις, συνθήκες για τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών για να βρει κανείς δουλειά. Uh, Ευχαριστώ για την ερώτηση. Σημαντική, βασικό. Θα μιλήσω στα Ολλανδικά, συγγνώμη. Uh, Νομίζω λοιπόν ότι αγγίζεται μια πάρα πολύ ευαίσθητη χορδή γιατί η δημιουργία θέσεων απασχόληση είναι κάτι παραπάνω από τη δουλειά από πλευρά των όσων αναζητούν θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει οργάνωση της εργασίας, να υπάρχει κινητικότητα, θα πρέπει να υπάρχει επαφή μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν συντονισμός από, και από τις δύο πλευρές και όπως ε, είπε ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ και όποιος έχει διαβάσει τις δηλώσεις του θα δει ότι το πρόγραμμα έχει να κάνει με τις θέσεις απασχόλησης αλλά και με την ανάπτυξη. Ανάπτυξη θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε και αυτός θα είναι στόχος της Επιτροπής αυτής για να υπάρξει ανάπτυξη και πιο πολλές ε, επενδύσεις. Δεν φτάνει η ανάπτυξη. Θα πρέπει η ανάπτυξη αυτή να σημαίνει και ανάπτυξη θέσεων εργασίας. Αλλά χρειαζόμαστε λοιπόν την ανάπτυξη αυτή. Ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 300 δισεκατομμύρια. Το έχουμε αναφέρει το ποσό αυτό. Υπάρχουν και πολλές πρωτοβουλίες που έχουν εξαγγελθεί για να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη στην έρευνα, στην καινοτομία μεταξύ άλλων. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχει υπερβολική ρύθμιση, να μην υπάρχουν τα νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια. Όλα αυτά θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο. Θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να υπάρξει πνεύμα επιχειρηματικότητας, να υπάρχει εμπιστοσύνη, να υπάρχει διάθεση για επενδύσεις. Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια αγορά κεφαλαίου προκειμένου να μην εξαρτώνται οι επενδυτές από τις τράπεζες, αλλά να μπορούν να προσφύγουν και στην αγορά. Και νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιτηρήσουμε σε μια ισορροπία προσφορά και ζήτηση. Και αυτό συνάδει και με την ε, κοινωνική οικονομία της αγοράς. Να υπάρχει λοιπόν ανάπτυξη και να υπάρχουν και θέσεις αποσχόλησης. Ε, να δώσω το λόγο στην Γιούτα Στάινλουκ που εκπροσωπεί τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Είχε το λόγο. Καλημέρα κυρία Τάισεν ε, και εξ ονόματος των σοσιαλδημοκρατών ε, σας καλωσορίζω σήμερα το πρωί. Οι άνθρωποι στην Ευρώπη αλλά και εμείς δικαίως αναμένουμε στην Ευρώπη να σταματήσει το κοινωνικό ντάμπινγκ και το ντάμπινγκ των μισθών, οι ανισότητες. Ε, όλα αυτά είναι η καθημερινότητα δυστυχώς για τους εργαζομένους. Ο πρόεδρος Γιούγκερ τάχθηκε υπέρ μιας ε, συνεπούς ε, ανάλυσης των αδυναμιών της αγοράς. Πού θεωρείτε εσείς όμως ότι ε, βρίσκονται τα συγκεκριμένα προβλήματα σε ό,τι αφορά την απόσπαση και συγκεκριμένα τι προτιθέστε να κάνετε για να βοηθήσετε και τους εργαζόμενους αλλά και τις οικονομίες, τις τοπικές σε ό,τι αφορά τον παράνομο ανταγωνισμό μισθών αλλά και τον παράνομο, τις παράνομες συνθήκες εργασίας. Πώς θα μας προστατεύσετε από αυτά. Ehm, Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά την απόσπαση των εργαζομένων είναι πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο και το γνωρίζουμε αυτό όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο τον τελευταίο καιρό, άλλωστε έχουμε δώσει πάρα πολύ προσοχή στο θέμα αυτό. Το σημαντικότερο που πρέπει να γίνει είναι ότι θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό πάντα. Έχει γίνει σχετική ανάλυση όπου έχουν εξεταστεί η οδηγία για τους αποσπασμένους, η βασική οδηγία για να δούμε μήπως πρέπει να αλλάξει. Και αυτή η τελική ανάλυση ελήφθησε η απόφαση ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να γίνει καλύτερη εφαρμογή, καλύτερη εκτέλεση. Γι' αυτό λοιπόν και υπήρξε εκτελεστική οδηγία. Θα πρέπει λοιπόν ε, αποτελεσματικά να εφαρμοστεί η οδηγία στα κράτη-μέλη. Τα νέα μέτρα που περιλαμβάνονται για την καταπολέμηση των καταχρήσεων θα πρέπει να γίνουν, να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικό τρόπο σε ό,τι αφορά και τις εποπτικές αρχές των εθνικών κρατών μελών. Μεγάλη προϋπόθεση και αυτή για την σωστή εφαρμογή. Και μετά θα πρέπει να εξετάσουμε το τι γίνεται στην πραγματικότητα, στην πράξη η οδηγία αυτή, εφαρμοστική οδηγία, όταν ε, τεθεί σε ισχύ και μετά από δύο χρόνια, αν δούμε ότι έχουμε επιλύσει κάποια από τα προβλήματα, ίσως όλα τα προβλήματα, εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι τότε θα πρέπει να γίνει να ληφθεί η απόφαση για το τι θα πρέπει να γίνει με την οδηγία αυτή. Αλλά στο μεταξύ δεν θα πρέπει να διστάζουμε, να εξετάζουμε και την οδηγία τη βασική οδηγία για την απόσπαση. Ξέρουμε ότι κάποιες βασικές ε, έννοιες όπως ε, η ελάχιστη μισθή παρουσιάζουν προβλήματα. Λοιπόν, αν υπάρχουν προβλήματα και ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, θα πρέπει να τολμούμε να ασκούμε κριτική και να ασχοληθούμε και με τη βασική οδηγία. Να δούμε κατά πόσο χρειάζεται μεταρρύθμιση, αλλά ξεκινήσουμε από την αρχή. Να εφαρμόσουμε την εφαρμοστική οδηγία, να δούμε τι θα αποφέρει να μην κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα εντωμεταξύ και να θέτουμε τα βασικά προβλήματα τα οποία περιλαμβάνονται στη βασική οδηγία. Αυτό εννοούσε και ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ όταν μίλησε για την στοχευμένη μεταρρύθμιση της οδηγίας για την απόσπαση. Ανθέα Μάκιντάιρ για το ECR. Ευχαριστώ. Κυρία Τάισεν, εδώ είμαι. Εκ μέρους της ομάδας του ΕΣΥΑΡ. χαίρομαι ιδιαίτερα σας βλέπω εδώ σήμερα το πρωί. Στο τέλος της προηγούμενης θητείας του Κοινοβουλίου υιοθετήσαμε μια έκθεση. Τίτλος της «Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία φιλόξενου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και για τις καινούριες επιχειρήσεις, για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης». Ήταν πρωτοβουλία της Επιτροπής Απασχόλησης. Τόνισε όλος ιδιαίτερος την πρόσφατη τάση Δηλαδή ότι οι εταιρείε επιστρέφουν την παραγωγή και τις υπηρεσίες τους στην Ευρώπη. Αυτό συνεπάγεται δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μοναδική ευκαιρία να επιταχύνουν αυτή την τάση της παλινόστησης και την επιστροφή των θέσεων απασχόλησης στα κράτη-μέλη. Συζητήσαμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία θηρίδα για να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις ε, εσείς πώς βλέπετε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε να επαναφέρουμε τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ κύριε Μάκιντάιρ. Θα πρέπει να φροντίσουμε σίγουρα να υπάρχει καλύτερο επιχειρηματικό κλίμα στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να υπάρξουν θέσεις απασχόλησης, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι θέσεις απασχόλησης και στον κρατικό τομέα, στο δημόσιο τομέα, αλλά αν θέλουμε επιπρόσθετες θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να είναι στο ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσει, θα πρέπει να, υπάρξει, ε, να υπάρξουν κίνητρα για να είναι ελκυστική η επένδυση από πλευρά των επενδύσεων, από πλευρά των επιχειρήσεων, θα πρέπει να έχουμε την τόλμη να δίνουμε να απασχολούμε άτομα, να δώσουμε ευκαιρίες για ανάπτυξη και όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα μέσο, ένας τύπος, μία μαγική λύση επί της οποίας θα επικεντρωθούμε. Όχι, είναι πολύ επίπεδο το πρόβλημα αυτό. Και όλα τα προσκόμματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτα και τα οποία εμποδίζουν την ανάπτυξη ή την δημιουργία, την ίδρυση επιχειρήσεων, όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αρθούν. Και νομίζω ότι μεταξύ άλλων ε, σε αυτά ασκεταλέγεται και η διοικητική απλούστευση. Και προ την κατεύθυνση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κρατήσει ένα ολόκληρο εργαλείο, ένα ολόκληρο μέσο, πάρα πολύ ωφέλιμο θεωρώ, για να... και θα πρέπει να αξιοποιηθεί πρωτού προβούμε σε περαιτέρω προτάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αλλά να γίνει και μια αξιολόγηση. Να γίνει μια αξιολόγηση των αποφάσεων που ήδη έχουμε λάβει. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει λοιπόν να τολμούμε να κάνουμε την άσκηση αυτή. Με ανοιχτό πνεύμα, με ανοιχτό όραμα και σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, ακόμα και την προστασία στον εργασιακό χώρο. Και ποτέ να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο απότερος σκοπός. Αυτό που προστατεύεται θα πρέπει να εξακολουθήσει να τη χάνει προστασία, αλλά θα πρέπει να κοιτάμε πώς μπορούμε ενδεχομένως να προσαρμόσουμε κανόνες προκειμένου να φροντίσουμε οι επιχειρήσεις και αυτές να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά χωρίς πάντα να χάνεται η διάσταση της προστασίας. Είχα κι άλλο να σας πω, αλλά δεν προωρώ μέσα σε δύο λεπτά να σας παρουσιάσω όλο το πανόραμα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει κάτι να γίνει για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα. Ιδάλλως δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης άλλες. Ευχαριστώ η Μάριαν Χάρκιν που εκπροσωπεί την Άλντε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι και σα καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Υποψήφια Επίτροπε. Είπατε στην κρατή σα απάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι μέχρι στιγμή αποτύχαμε στην υλοποίηση πολλών στόχων τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020. Και αυτό ισχύει σε ό,τι αφορά το στόχο κοινωνικού αποκλεισμού και τη μείωση τη ανεργία. Και μάλιστα είπατε πριν από λίγο ότι ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ είπε ότι θα πρέπει να σταθμίζουμε τι κοινωνικέ επιπτώσει όλων των μέτρων που υιοθετούμε. Δεδομένων των επιτευγμάτων για του στόχου του 2020 και της αλληλεξάρτησής τους με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τι αλλαγές χρειάζονται κατά τη γνώμη σας στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο προκειμένου να υλοποιήσουμε τους στόχους μας για το 2020, δηλαδή να περιλάβουμε περισσότερους κοινωνικούς δείκτες, να ενισχύσουμε την εφαρμογή τους και να εξασφαλίσουμε ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία ή ενδεχομένως οποιαδήποτε άλλη πρόταση έχετε εσείς να κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, όντω, αυτά τα δύο συνδέονται το ένα με το άλλο και θα πρέπει να φροντίσουμε και το ευρωπαϊκό εξάμεινο να καταστεί πιο κοινωνικό. Αυτό προκύπτει από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Προέδρου Γιούγκερ. Αυτή είναι η εντολή που λάβαμε και εγώ ιδιαίτερα στο χαρτοφυλάκιό μου. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν στο εξάμεινο για να τονίσουμε τους στόχους του 2020, για να καταστήσουμε το εξάμεινο πιο κοινωνικό. Έχουμε διάφορες δυνατότητες, αλλά και καθήκοντα θα έλεγα, στην επόμενη περίοδο. Καταρχάς, οι κοινωνικοί δείκτες. Υπάρχουν κοινωνικοί δείκτες, αλλά ε, αντιμετωπίζονται με κάπως ε, ε, δευτερεύοντα ρόλο. Είναι βοηθητικοί μόνο. Τους εξετάζουμε αλλά δεν τους χρησιμοποιούμε. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε μια προσπάθεια. Και αυτή είναι η συμφωνία άλλωστε εντό της ομάδας των μελλοντικών επιτρόπων να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στους κοινωνικούς δείκτες και επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να τους υπαγάγουμε στο ίδιο επίπεδο όπως οι δείκτες για τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισοτήτων. Από τη στιγμή δηλαδή που εντοπίσουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, να γίνεται μία ανάλυση εις βάθος, προκειμένου να έχουμε πολύ καλύτερη γνώση του τι συμβαίνει στα κρατημέλη. Και αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί και στις συστάσεις αναχώρα. Κάτι άλλο που θα πρέπει να γίνει. Δεύτερο στοιχείο θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην διαδικασία αυτή και οι κοινωνικοί εταίροι. Γιατί γίνονται πολλές συστάσεις. Συστάσει σε τομεί όπου είναι αρμόδια τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα επιρροή, Θα πρέπει να κάνουμε πιο πολλέ συστάσει, αλλά και διαφορετικέ συστάσει. Από πλευρά όμω κρατών μελών υπάρχει αντιμετώπιση ότι α, γιατί ανακατεύεται η Ευρώπη με τα δικά μα, Θα πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθούν καλύτερα τα κοινοβούλια. Νομίζω ότι αν γίνει αυτή η άσκηση, αυτή πριν καταρτιστούν οι αιτήσεις Επισκόπηση ανάπτυξης, θα πρέπει να συμπεριληφθεί λοιπόν το κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το μεκρονοϊκό διάλογο, τι συστάσεις αναχώρα. Όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν και θα πρέπει να ακούσουμε με προσοχή ο ένας τον άλλον προκειμένου να διαμορφώσουμε πραγματικά με το βέλτιστο δυνατό τρόπο αυτό το εργαλείο. Ευχαριστώ. Ειρήνα Ρόνια Κάρη από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κυρία Τάισεν. Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή που μας κάνατε. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στις βασικές προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Βλέπουμε όλο και περισσότερο την πίεση που υφίστανται οι άνεργοι να αυτοαπασχοληθούν και την προσπάθεια των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να αποφύγουν ε, την πληρωμή αδειών ε, μητρότητας ε, και ούτω καθεξής. Υπάρχει τεράστια πίεση λοιπόν και οι πιλότες, και οι πιλότες συγγνώμη, δηλώνουν ότι αισθάνονται μεγάλη πίεση και αυτό επηρεάζει και τις επιδόσεις τους. Τι θα κάνετε προκειμένου να ελαφρύνετε αυτή την πίεση των αυτοαπασχολούμενων, τι ε, μέτρα θα λάβετε ώστε να εξασφαλιστούν και κατάλληλες συνθήκες για το προσωπικό πτήσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Αυτό το πρόβλημα του απασχολούμενου είναι πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα, ένας γορτίος δεσμός, μια ε, παράνομη ουσιαστικά χρήση των εργαζομένων. Ποιοι θα πρέπει λοιπόν να αντιδράσουν, καταρχάς τα κράτη-μέλη, να φροντίσουν να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες που θέτουν. Σίγουρα στην κοινωνία υπάρχουν ε, χώροι όπου ασκείται πίεση στον κόσμο να εργαστεί ως αυταπασχολούμενος. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό. Δεν έχει ε, επιλογή ο κόσμος να αποφασίσει αν θα είναι αυτοαπασχολούμενος ή μισθωτός. Υπάρχουν κανόνες. Αν ε, λοιπόν δεν είναι στο χέρι του εργαζόμενου να αποφασίσει, θα πρέπει λοιπόν από πλευρά Ευρώπη έχουμε εμεί σίγουρα, γιατί το πρόβλημα αυτό είναι και διασυνοριακό. Αλλά επιπλέον, όταν υπάρχει ο κόσμος ο οποίος ε, παρανόμως παρουσιάζεται ως αυτοπασχολούμενος, αυτό τι σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται και η νομοθεσία που έχουμε θέσει εμείς από ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα ωραία εργασία, σε ό,τι αφορά ε, τα επιδόματα εγκυμοσύνης. Δεν γίνονται σεβαστοί λοιπόν οι κανόνες μας. Είναι απάτη αυτό και θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα στην Ευρώπη ε, σε ό,τι αφορά τη μαύρη εργασία εδώ λοιπόν εμπίπτει το θέμα αυτό και είμαι πεπισμένη ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερε προσπάθειε για να συλλέξουμε πιο πολλά στοιχεία από τα κράτη-μέλη, να σχηματίσουμε μια καλή εικόνα για του ε, ψευτοαπασχολούμενου και να δούμε πώ και εμεί από δική μα πλευρά μπορούμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίε για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό. Αλλά είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το ζήτημα αυτό. Και θα υποστηρίξω όσους θέλουν να το καταπολεμήσουν άλλωστε. Thank you. Ευχαριστώ. Η Τζιν Λάμπερτ από τους Πρασίνους έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθες Αντάισεν εκ μέρους της ομάδας μας επίσης. Και εγώ θέλω να αναφερθώ στη δημιουργία θέσεων εργασίας και σε αυτά που έλεγες ότι θες μια βιώσιμη Ευρώπη. Διότι από την άποψη των ε, Πρασίνων τα καθήκοντα που σας ανέθεσε ο κύριος Γιούνκερ δεν δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης μέσω πρασινίσματος της οικονομίας και κεφαλοποίησης ε, μιας πράσινης μετάβασης όσον αφορά τα επιδόματα. Ε, εσύ τι θα έκανες για να προωθήσεις τις πράσινες δεξιότητες το όλο πρόγραμμα της πράσινης μετάβασης στην Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως όσον αφορά το πακέτο για επενδύσεις, θέσεις απασχόλησης και για ανάπτυξη. Μήπως υπάρχουν τρία συγκεκριμένα βήματα στα οποία θα έθετες προτεραιότητα στο συγκεκριμένο τομέα. Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά τις πράσινες θέσεις εργασίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθεί προσοχή στην κρίση τι είδαμε, ότι χάσαμε πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε αφελείς και να πιστεύουμε ότι θα ξαναδούμε και θα ξαναβρούμε τις ίδιες θέσεις εργασίας. Είναι σε μετάβαση, σε μεταβατική φάση και η οικονομία και η κοινωνία μας. Έχουμε πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά τους πόρους μας, σε ό,τι αφορά την ενέργειά μας, σε ό,τι αφορά τον άνθρακα και χρειαζόμαστε πιο πολύ βιωσιμότητα. Άρα αυτό θα πρέπει να είναι η βασική κατεύθυνση και η κατευθυντήρια γραμμή μας, ο μύτος όλων των πολιτικών μας. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μεταφραστεί και σε ό,τι αφορά την πολιτική για τη θέση της απασχόλησης. Θα πρέπει η μετάβαση αυτή να γίνει δυνατή και στην αγορά εργασίας. Ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στη θέση εργασίας, σε, στην αγορά εργασίας ή όσοι έχουν χάσει τη θέση εργασία τους ή οι νέοι που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να δουλεύουν, θα πρέπει όλοι να έχουν τις σωστές ικανότητες για να μπορούν να τοποθετηθούν στους νέους τομείς, στις νέες επιχειρήσεις. Αυτό θα πρέπει να το φροντίσουμε, θα πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια και από πλευρά κατάρτιση, εκπαίδευση, να υπάρχουν οι σωστέ και οι απαραίτητε ικανότητε, τα σωστά προσόντα. Υπάρχουν πρωτοβουλίε για πράσινε επιχειρήσει, για πράσινε θέσει απασχόληση, για κυκλική οικονομία. Όλα αυτά θα πρέπει να προωθηθούν. Δεν είναι κάτι περιθωριακό αυτό, αλλά κάτι πολύ βασικό για μια κοινωνία σε μεταβατική φάση. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, θα πρέπει να τολμήσουμε να επενδύσουμε σε καινοτόμα έργα, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για πειραματισμούς και θα πρέπει να τολμήσουμε να χρησιμοποιήσουμε όσα μέσα έχουμε στη διάθεσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you. Σας ευχαριστώ. Λάωρα Αγκέα από το EFTD. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Αξιότιμη κυρία Τάισεν, γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε κάποιες χώρες ε, υπάρχει το εισόδημα το κειμένων που επιτρέψει εκείνο που δεν βρίσκει και μια απασχόληση να ζει με αξιοπρεπή τρόπο. Ενώ περιμένει να βρει μια καινούρια δουλειά. Εν τω μεταξύ έχει τη δυνατότητα υπό μορφή κοινωνικών ε, εργασιών επιστρέψει αυτά που λαμβάνει. Αυτό το μέσο είναι αποτελεσματικότατο σταθεροποιητή των αρνητικών συνεπειών της κρίσεως και των πολιτικών λιτότητας που ζει εδώ και πολύ χρόνο η Ευρώπη σε αυτά τα μέρη. Θα συστήνατε όλες οι χώρες να αναλάβουν την υποχρέωση να εγγυηθούν το εισόδημα των, ε, της υπηκότητας στους πολίτες και πιστεύετε ότι είναι θεμελιώδη σημασία σε τέτοιες δύσκολες και ευαίσθητες στιγμές που ζούμε. Θα ήθελα ε, να σας αναθέσω το καθήκον να, να επιστρέψετε την εμπιστοσύνη στους ε, πολίτες, διότι δεν δίνονται τα απαραίτητες εγγυήσεις στους πολίτες και δεν έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ελάχιστο μισθός για την επιβίωση, ένα ελάχιστο εισόδημα για τον κόσμο. Η προσωπική μου άποψη για αυτό είναι ότι στον 21ο αιώνα αυτό πρέπει να μπορούμε να το παρέχουμε στον κόσμο και σε επίπεδο κοινωνίας θα πρέπει να παροτρύνουμε στον κόσμο σε όσους μπορούν αλλά και όσους δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγους θα πρέπει να τους βοηθήσουμε, να τους προστατεύσουμε, να τους δώσουμε ένα ελάχιστο εισόδημα. Πολύ βασικό εργαλείο. Αν λοιπόν αποφάσιζα εγώ, σε όλα τα κράτη-μέλη θα υπήρχε ελάχιστος μισθός. Αλλά, αλλά, δεν έχουμε την ερμοδιότητα από πλευράς Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν μια συνθήκη και κανόνες που θα πρέπει να σεβαστούμε. Από πλευράς Ευρώπης λοιπόν μπορούμε να δώσουμε κίνητρα δεν μπορούμε όμως να επιβάλλουμε τίποτα. Αυτό αφενός. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα και το κάνουμε αυτό έμεσα με διάφορες συστάσεις αναχώρα, όπου για παράδειγμα εξετάμε πώς ε, μπορούμε να οργανώσουμε την καταπολέμηση της φτώχειας και της κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό είναι ένα μέσο, αλλά δεν αρκεί προφανώς. Δεν αρκεί με ένα ελάχιστο εισόδημα, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι άνθρωποι αυτοί, να υπάρξει επένδυση στον άνθρωπο, να έχουν μια ευκαιρία να βγουν από τη φτώχεια και να ξαναξεκινήσουν, να δουλεύουν, να τους καθοδηγήσουμε προς την αγορά εργασίας. Και αν το εξετάσουμε αυτό αποκινούμε το ελάχιστο μισθό, θα πρέπει να φροντίσουμε αυτός ο ελάχιστος μισθός σε, κάθε χώρα να μην γίνει ένα δίκτυο ασφαλείας, στο οποίο τελικά θα παγιδεύεται ε, το άτομο. Θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή ισορροπία μεταξύ της διάθεσης του μισθού αυτού και των κινήτρων αφετέρου που χρειάζονται προκειμένου να καθοδηγείται ο κόσμος στον φυσιολογικό κύκλο της εργασίας. Μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την ε, υποστήριξη των κρατών μελών για να υπάρχει ένα, ένας προϋπολογισμός αναφοράς. Αλλά αυτό μπορούμε μόνο να το συστήσουμε, δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Ε, Ευχαριστώ ο κύριος Φουντούλης από τους μη εγγεγραμμένους. Και αν τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα παρακαλώ. Δύο σημαντικά θέματα θα ήθελα να θέσω υπόψη σας και θεωρώ πως θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη απάντηση εκ μέρου σας. Πρώτον, ποιες συγκεκριμένες νομοθετικές και μη πρωτοβουλίες θα αναλάβετε ώστε να διασφαλιστεί ένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων με ειδικέ ανάγκες και των ατόμων με αναπηρία. Γνωρίζετε κι εσείς όπως όλοι μας πως τα άτομα αυτά είναι τα μεγαλύτερα θύματα της οικονομικής κρίσης. Στη χώρα μου την Ελλάδα, πολλά άτομα με αναπηρία δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακα και σε στοιχειώδη ιατρική και νοσοκομιακή περίθαλψη. Να μην αναφερθώ και στο ότι τα άτομα με νοητική υστέρηση έχουν αποκλειστεί και από τα προγράμματα της διαβίου μάθησης. Τι θέλουν λοιπόν οι συνάνθρωποι μας αυτοί, εκπαίδευση, εργασία και περίθαλψη. Δεύτερον, μιλάτε συνεχώ για την ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και την κινητικότητα έχετε λάβει υπόψη σας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει μαζική εσωτερική μετανάστευση, μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες όπως τη δική μου την Ελλάδα και τις χώρες του Νότου. Οι νέοι επιστήμονες και τα καλύτερα μυαλά της χώρας να αναζητούν σε άλλες χώρες ευκαιρίες για εργασία. Η ανάπτυξη που όλοι περιμένουμε πώς μπορεί να έρθει σε μια χώρα στην οποία οι νέοι να βρουν τα μέσα και τον τρόπο για να φύγουν από ευχαριστώ. Eh, Uh, Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Πολλές ερωτήσεις μαζεμένες θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες συνοπτικά. Τι μπορούμε να κάνουμε για τους ανάπηρους, για τα άτομα με ε, περιορισμούς. Καταρχάς λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία διαφορετική εικόνα. Και εδώ θα ήθελα να συνδράμω. Τα άτομα με περιορισμούς είναι και άτομα με ταλέντα. Είναι άτομα με ικανότητες. Και όχι επειδή έχουμε κάποιους περιορισμούς σε κάποιους τομές ή με το άτομο αυτό περιορισμένο γενικότερα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να σεβαστούμε την νομοθεσία που ήδη υφίσταται για να μην υπάρχουν διακριτικέ μεταχειρήσει στην αγορά εργασία. Υπάρχουν κάποιε προνομιακέ μεταχειρήσει για τα αναπηρά άτομα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασία. Θα πρέπει να γίνονται σεβαστά λοιπόν αυτά. Και θα πρέπει να το φροντίσουμε αυτό. Επίση, υπογράψαμε μία συνθήκη του ΟΗΕ για τα ανάπηρα άτομα που ε, προσδίδει κάποια θεμελιώδη δικαιώματα στα ανάπηρα άτομα. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν όλα αυτά αποτελεσματικά να εφαρμοστούν. Και πολύ συγκεκριμένα πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι βραχυπρόθεσμα. Θα πρέπει να αναλάβουμε και ε, νομοθετικό έργο ενδεχομένως για να υπάρχει μεγαλύτερη προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Υπήρξε τέτοιο αίτημα και από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρω ότι οι υπηρεσίε εργάζονται για να υποβάλουν μια πρόταση οδηγίας προκειμένου να φροντίσουν ότι θα δημιουργηθεί μια πραγματική ενιαία αγορά για προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία προκειμένου να είναι πιο προσβάσιμα, να είναι πιο φθηνά τα προϊόντα αυτά και οι υπηρεσίες αυτές και η ενιαία αγορά να μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα και για τους αναπήρους. Τι θα κάνουμε με την κινητικότητα τώρα κατά πόσον αυτό συνδράμει στις μεταναστευτικές ε, ροές. Ίσως. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές ε, ε, πάρα πολλά παραδείγματα και θεωρώ ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την εργασιακή κινητικότητα γιατί αυτό και για την μικροοικονομία είναι καλό αλλά και για την μακροοικονομία. Και θα ήθελα να αναπτύξω περαιτέρω αυτό το θέμα αυτό σε κάποια επερχόμενη ερώτηση ενδεχομένω. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το ξεχάσουμε αυτό, γιατί γενικά συνολικά η κινητικότητα είναι κάτι θετικό στην Ευρώπη και θα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Thomas Mann. Ευχαριστώ. Thomas. Ο Τόμας Μαν από το ΕΛΚ. Κυρία υποψήφια, αγαπητή Μαριάννε, επί 20 χρόνια ήσουν μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχεις αποδείξει επανειλημμένα πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να είναι αισθητή στα 5 εκατομμύρια νέους άνοργους. Έχουμε θέσει ένα μήνυμα. Θέλουμε να μειωθεί η ανεργία των νέων. Υπάρχουν και μέσα όπως ε, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση. Αυτά τα έχει θέσει και ο Πρόεδρος Γιούγκερ. Τι μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε από την Επίτροπο Τάισεν προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρω το δυναμικό τη πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και τι μπορεί να κάνουμε για τα κράτη-μέλη προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν εκχωρηθεί, δεν γίνεται σωστή κατανομή, πού είναι τα προβλήματα ή μήπως λείπει η προθυμία για να δράσουμε. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη. Eh, ε, σας ευχαριστώ, συνάδελφε Μαν. Μιλώντας για την ανεργία των νέων, από πλευράς Ευρώπης ε, σκεφτόμαστε τα 5,7 εκατομμύρια νέους που δεν έχουν ε, θέσεις απασχόλησης τα 7 εκατομμύρια νέους που δεν έχουν καν και θέση κατάρτισης. κοιτώντα όμως και την πρωτοβουλία για τους νέους, όπου δημιουργήσαμε ένα χρηματοοικονομικό πλαίσιο και αναρωτιόμαστε γιατί δεν χρησιμοποιούνται οι δαπάνε αυτές, τα κονδύλια αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα για τις εγγύησεις για την νεολαία, από τα προγράμματα και τις δεσμεύσεις των κρατών μελών για να φροντίσουν να διοχετευτούν οι νέοι προς την αγορά εργασίας και να φροντίσουν μέσα στους τρεις-τέσσερις μήνες που ε, έπονται μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης να βρεθούν είτε σε μια θέση απασχόλησης είτε σε μια θέση κατάρτισης. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε. Λαμβάνονται μέτρα ακόμα και κράτη-μέλη που δεν χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τους νέους θα πρέπει να λάβουν σχετικά μέτρα προκειμένου να υπάρχει μετάβαση των νέων αυτών από την, τις σχολές ή από την ανεργία στην εργασία. Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για τους νέους θα πρέπει να την προωθήσουμε και απο ευρωπαικη πλευρά πλευράς έχει γίνει ένα front-loading όλων των δαπανών. και έχουν γίνει προσπάθειες για κάποια κρατημέλη να θέσουν σε λειτουργικότητα τα προγράμματα ήδη μέχρι τα τέλη του 2014. Αυτό το έχουν κάνει κάποια κρατημέλη, κάποια άλλα όχι. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνονται σεμινάρια, δίνονται κατευθυντήριε γραμμέ προκειμένου να υποστηριχθούν τα κρατημέλη. Προκειμένου να δουν τα κρατημέλη πώ μπορούν να καταρτήσουν προγράμματα τα οποία γρήγορα να μπορούν να τα εφαρμόσουν πέρα από τα διοικητικά προβλήματα και κλείνει το μικρόφωνο τη ομιλητρία. Ο Σον Σάιμον από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ. Για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Ο πρόεδρος Γιούγκερ υποσχέθηκε μία αναθεώρηση εδώ και τώρα τις οδηγίες για τους ε, αποσπασμένους εργαζόμενους και όχι μία όριστη χρονική στιγμή στο μέλλον. Εσείς όμως ήσταν αρκετά ασαφείς. Μιλήσατε εκτενώς για την ε, οδηγία της ε, εφαρμογής, αλλά η νομολογία Ράκιν Λαβάλ υπονόμευσε τη νομική βάση της αρχικής οδηγίας. Αυτή η αρχική οδηγία χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ρητά και κατηγορηματικά. Ήδη αθετείτε την υπόσχεση του Πρόεδρου Γιούγκερ για ριζική αναθεώρηση αρχικής οδηγίας. Ε, αυτό σημαίνει ότι διαφωνείτε μαζί του. Αν όμως θέλετε να τηρήσετε την υπόσχεση του, τι εννοείται στοχοθετημένη αναθεώρηση. Χρειαζόμαστε μία ριζική αναθεώρηση και όχι μία απλή επανεξέταση. Αλλιώς αυτό θα είναι ένα παραπέτασμα καπνού. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή γιατί μου επιτρέπει να κάνω περαιτέρω διευκρινήσεις στο θέμα αυτό. Έχουμε εγκρίνει μία εφαρμοστική οδηγία η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο. Να εφαρμοστεί για να δούμε κατά πόσον θα ε, επιφέρει τις βελτιώσεις που επιθυμούμε, δηλαδή η απόσπαση να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε συμφωνήσει. Αυτό αφενός. Κατά δεύτερον, θα γίνει μια αξιολόγηση και θα δούμε κατά πόσον χρειάζεται κάτι παραπάνω να γίνει. Σε ό,τι αφορά την βασική οδηγία του 96 και αυτή θα πρέπει να τολμήσουμε να την εξετάσουμε στο μεταξύ. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο κανόνας, κατά πόσον εφαρμόζεται αν εφαρμόζονται ή αν δεν εφαρμόζονται, τι μπορούμε να κάνουμε για να την εφαρμόσουμε καλύτερα. Σε περίπτωση που ο κανόνας δεν είναι καλός, θα πρέπει να τον βελτιώσουμε. Πάντα θα πρέπει να γίνεται μια ανάλυση, μια αξιολόγηση βάσει στοιχείων, δεδομένων και βάσει της καλής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Να δούμε κατά πόσο μια τέτοια οδηγία θα χρειαστεί να την αναθεωρήσουμε ή όχι. Και αυτός θα είναι ο τρόπος που θα εργαστώ. Δεν έχω πρόβλημα για την αναθεώρηση, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι το κουτί της Πανδώρας και ότι είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό. Σύμφωνοι. Θα πρέπει να δούμε κάποια τμήματα, αν χρήζουν τροποποίησης ή όχι. Αλλά η αρχή της απόσπασης είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβήτα το γεγονός ότι υπάρχει κόσμος, ότι υπάρχει η ελευθερία παροχής υπηρεσιών και ότι υπάρχουν ε, άνθρωποι που είναι αποσπασμένοι σε άλλα κρατημέλη, αυτή είναι μια αρχή που θέλω να κρατήσω. Πουθενά δεν αμφισβητείται αυτό. Ούτε από τον πρόεδρο Ζαν Jean-Claude Juncker, Όταν λέμε στοχθετημένη αναθεώρηση, αυτό τι σημαίνει να δούμε κατά πόσο υπάρχουν προβλήματα και αν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά μέσω αλλαγή της νομοθεσίας εφόσον ενδείκνεται αλλά σε πρώτη φάση περαιτέρω αξιολόγηση. Εφαρμογή, να δούμε πού βρισκόμαστε, ε, στο μεταξύ να γίνει αξιολόγηση και εφόσον είναι απαραίτητο, μεταρρύθμιση να θεώρησε τις οδηγίες του 96. Ε, ο κύριος Αρνεγκέρικε, συγγνώμη, από τους μεταρρυθμιστές και συντηρητικούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, βιώσιμη δημογραφική, δημογραφική ανάπτυξη. Μπορείτε να συντονίσετε καλύτερα την οικογενειακή πολιτική σε ό,τι αφορά την διακριτική μεταχείριση των οικογενειών με παιδιά στην ενιαία αγορά. Θα ταχθείτε υπέρ αυτών. Θα ταχθείτε υπέρ μια συνεπούς ε, πολιτικής υπέρ των ευρωπαϊκών οικογενειών που θα είναι και υπέρ του συμφέροντος του Ζαν Κλοντ Γιούγκερ αυτό μιλάτε για κοινωνική προστασία. Υποστηρίζετε τη γύρανση της Ευρώπης μέσω μιας αλλαγής κουλτούρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η άποψή σας για την κατάπληψη στον χώρο εργασίας και τι σκοπεύετε να κάνετε στη σχετική οδηγία. Θεωρείτε ότι η προστασία της εργασίας ό,τι αφορά τις Κυριακές αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οδηγίας αυτής και αν όχι γιατί. Σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις που μου θέσατε. Θα προσπαθήσω να δώσω μία απάντηση στις περισσότερες ε, εξ αυτών. Για την οικογενειακή πολιτική. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα των κρατών μελών, αλλά θα πρέπει να ασκούμε πολιτική που θα επιτρέπει στα κρατημέλη να ασκεί την πολιτική υπέρ των οικογενειών. Θα πρέπει να δώσουμε περιθώριο και να δώσουμε και κινήτρα όπου είναι αυτό δυνατόν. Ξέρετε όλοι ότι όταν μιλάμε για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, για προσόντα και κατάρτιση των ατόμων, όλα αυτά ξεκινούν στην οικογένεια, στις ευκαιρίες που δίνουν στα παιδιά από τη στιγμή που γεννιούνται. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις οικογένειες, θα πρέπει να υποστηρίζουμε τις οικογένειες, τα παιδιά, τη φύλαξη, να υπάρχει κατάρτιση, εκπαίδευση. Και θα πρέπει όλα αυτά να μας απασχολήσουν. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ εργασία και οικογένεια. Και αυτό το κάνουμε μέσω τη νομοθεσία για τα εργασιακά. Όσοι δουλεύουν θα πρέπει να έχουν και χρόνο για να εκτελέσουν τα οικογενειακά του καθήκοντα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σχετική εργασιακή νομοθεσία. Τι κάνουμε για του ε, πρεσβύτερου, για του ηλικιωμένου στην αγορά εργασία. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει καταρχά να φροντίσουμε να απασχολούνται, να είναι ενεργοί και δραστήριοι οι ηλικιωμένοι. Τους χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην κατάρτιση διαβίου, στην ε, κατάρτιση ενηλίκων. Πολύ σημαντικό αυτό για να διατηρηθούν ενεργοί οι άνθρωποι αυτοί όσο θέλουν και όσο μπορούν να μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά εργασία. Το χρειάζονται. Και θέλουμε να αυξήσουμε και τα όρια συνταξιοδότησης, την ηλικία συνταξιοδότησης, να μπορεί να εργάζεται ο κόσμος όσο το επιθυμεί και επίσης όταν φτάνει σε ηλικία συνταξιοδότησης να έχει μία αξιοπρεπή σύνταξη, να κάνουμε όλες τις προσπάθειες που συμφωνήσαμε και που περιλαμβάνονται και στις συστάσεις ανά χώρα για να διαμορφωθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα συνταξιοδοτικά μας ε, συστήματα. Η κυρία Μπέτρις Μπεσέρα από τους Φιλελεύθερους. Καλημέρα σας κυρία Τέισεν. Εδώ είμαι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα θέλησε να είπε ότι θα αποσύρει την οδηγία του 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε μπλοκάρει το Συμβούλιο για την άδεια μητρότητα. Σε αυτήν την τετραετία η αρχή κρατών και κυβερνήσεων είπε διάφορα ωραία λόγια, αλλά υπάρχει παρόλα αυτά ανασχετική μειοψηφία εμείς τα κοινοτικά θεσμικά όργανα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κατάλληλη κάλυψη στους εργαζομένους όταν δεν μπορούν ε, να εργαστούν. Όπως ε, συμβαίνει με τις ε, γυναίκες πριν τον τοκετό. Δικαιούνται άδεια μητρότητας. Θα πρέπει να συμφιλιώσουμε τον οικογενειακό βίο με τον επαγγελματικό. Δεν θα πρέπει να θεωρείται πολυτέλεια το να αποκτήσει κανείς παιδί. Δεν θα πρέπει επουδενή φυσικά να ξεχάσουμε το γενικό συμφέρον, δηλαδή το συμφέρον των 500 εκατομμυρίων συμπολιτών μας, όχι των συμφέροντων μιας χώρας ή μιας κυβέρνησης. Ε, το 2010 ήταν υπέρ της διεύρυνσης της άδειας μητρότητας. Λυπούμε, αλλά η πρόεδρος διέκοψε την κυρία Μπεσέρα. Μου επιτρέπετε να υποβάλω την ερώτησή μου, κυρία Πρόεδρε. Ήδη έχουμε ένα δεκάλεπτο καθυστέρηση. Δηλαδή, θα στερήσουμε από πέντε ομιλητέ ε, την δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις. Νομίζω ότι η κυρία Τέισεν σας κατάλαβε. Κατάλαβε τι ερώτηση θέλατε να υποβάλλετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά την άδεια μητρότητας, ε, ε, τα επιδόματα μητρότητα. φυσικά όλα αυτά είναι και εκτιμένα δικαιώματα, δεν πρόκειται να τα αγγίξουμε και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Συμφωνία που υπάρχει για την ελάχιστη προστασία αυτό αποτέλεσε επιθυμία διαφόρων παραγόντων να αυξηθούν όλες αυτές αυτά τα επιδόματα. Αυτό προκάλεσε ε, ταραχή στο Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο υπήρξε συμφωνία και, και εγώ πιστεύω ότι τα επιδόματα μητρότητας είναι απαραίτητα. Και θεωρώ ότι στον 21ο αιώνα, όταν μιλάμε για την υγεία της μητέρας και του παιδιού, θα πρέπει να είναι απαράβατα τα θέματα αυτά, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και τους πατέρες, θα πρέπει να παροτρύνουμε και τους πατέρες να αναλάβουν τμήμα της φροντίδας αυτής. Γιατί αυτό είναι καθοριστικό και για τις περαιτέρω ευκαιρίες που θα έχει η οικογένεια, για τις ευκαιρίες που θα έχει η μητέρα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην κοινωνία και στην εργασία. Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες λοιπόν για να διαιρεθεί αυτή η φροντίδα. Και αν μπορούμε να φροντίσουμε να το βοηθήσουμε αυτό από πλευρά Ευρώπη, θα πρέπει να το κάνουμε. Τώρα, για το θέμα το άλλο θα πρέπει να μιλήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εμείς ε, στο Κοινοβούλιο είχαμε προτείνει τις 20 εβδομάδες, 22 εβδομάδες. Αυτό ήταν ε, υπερβολικά μεγάλο διάστημα για το Συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα εφικτό βήμα προς τα εμπρός. Θα πρέπει να το θέσουμε επιτάπητος. Θα πρέπει να το συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορεί να συμπεριληφθεί αυτό ως άδεια και ως ε, σύστημα φροντίδας για τους πατέρες κατά πόσον μπορεί να κατοχυρεθεί αυτό στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κυρία Επίτροπε, ψηφία Επίτροπε, απαριθμίσατε προτεραιότητες, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου. Συμφωνείτε να ξεκινήσει μια πρωτότυπη δουλειά μεταξύ της Επιτροπής Απασχόλησης μαζί σας και με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων που εδώ και ένα χρόνο πρότεινε ένα σχέδιο για επενδύσεις, για βιώσιμη ανάπτυξη και για ποιοτική απασχόληση κινητοποιώντας την αξία περίπου του 2% του πλούτου που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για νέα επενδυτικά σχέδια, για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που είναι απαραίτητε, ούτω ώστε μακροπρόθεσμα να δημιουργηθούν 10 εκατομμύρια θέσεις απασχόληση. Θα συμφωνούσατε να κινηθείτε προ αυτή την κατεύθυνση. Αξιότιμε συνάδελφε, θα πρέπει να ομολογήσω με πάσα ειλικρίνεια ότι θα πρέπει να ενημερωθώ για το σχέδιο αυτό, αλλά μπορώ να σα διαβεβαιώσω στην παρούσα φάση ότι είμαι διατεθειμένη να αναπτύξω μια σωστή και καλή σχέση με του κοινωνικού εταίρου. Ξέρω ότι οι κοινωνικοί εταίροι δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι. Ο κοινωνικό διάλογο δεν βρίσκεται στην καλύτερη φάση, στο καλύτερο επίπεδο απόδοση. Πέρασε μια σοβαρή κρίση το οποίο και δυσκολεύει και τους κοινωνικούς εταίρους να αποδεχτούν σε λύσεις. Το κατανοώ αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να ξαναξεκινήσουμε από κοινού με τον συνάδελφο τον που είναι υπεύθυνο για τον κοινωνικό διάλογο, τον Αντιπρόεδρο και μαζί με όλους τους επιτρόπους θα πρέπει να ακούσουμε και τους εκπροσώπους ε, ε, των ε, εργοδοτών αλλά και για τους εκπροσώπους της ΕΤΟΚ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη συμπερίληψη των κοινωνικών εταίρων, να είστε σίγουρος ότι θα είμαι σύμμαχός σας. Και θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί μπορούν να βοηθήσουν να γνωρίζουμε καλύτερα τις συνθήκες, γιατί αυτοί βρίσκονται επί τόπου κάθε μέρα και αυτοί μπορούν να φροντίσουν να λαμβάνουμε από κοινού αποφάσεις οι οποίες να έχουν καλύτερη αποδοχή, καλύτερη σύνδεση με την αγορά εργασίας και ξέρουμε ότι αν υπάρχει καλύτερη αποδοχή από τον κόσμο των αποφάσεων αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Άρα σε ό,τι αφορά το κατά πόσο ε, θα ακούσουμε τους κοινωνικού εταίρους, κατά πόσο θα συμμετέχουν, κατά πόσο θα διαβουλευτούμε μαζί τους, σίγουρα να με θεωρείτε σύμμαχό σας. Ευχαριστώ, Lambert, από Κυρία Τάισεν, είπατε εισαγωγικά ότι το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η οικονομική και η κοινωνική διακυβέρνηση προχωρούν παράλληλα και χρειάζεται ισότιμη αντιμετώπιση. Και ο πρόεδρος Γιούνκερ το αναφέρει αυτό. Ανησυχούμε όμως πολύ από μας. Η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή τίνει να επιβάλλει την ε, κυριαρχία της οικονομικής διακυβέρνησης. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα έχετε τη δύναμη να εξετάζετε τις προτάσεις που έρχονται από άλλους φορείς Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ίσως τελικά να αύξαναν την φτώχεια και την ισότητα και άρα θα αντέβαιναν τους στόχους ε, του 2020 για την μείωση της φτώχειας. Αν αυτό πιστεύετε, πώς μπορείτε να σταματήσετε να αλλάξετε αυτές τις προτάσεις που εμπεριέχουν τους κινδύνους. Έχετε και τη δυνατότητα να προβάλλετε βέτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το οικονομική διάσταση σε ό,τι αφορά την κοινωνική και οικονομική διακυβέρνηση. Νομίζω ότι υπάρχει σαφής αναφορά στις κατευθυντήριες γραμμές σε ό,τι αφορά και τις εντολές που λάβαμε από τον Ζαν Κλοντ Γιούγκερ στην ε, σχετική δήλωση αποστολής. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν κοινωνικά να υπάρχει, να υπάρχει μεγαλύτερη, ε, να υπάρχει μεγαλύτερη, μεγαλύτερο βάρος στην κοινωνική διάσταση σε ό,τι αφορά το κατά πόσον έχω δικαίωμα βέτο. Εργαζόμαστε ως ομάδα. Αυτή είναι η πρόθεση όλων των επιτρόπων. Όλοι να λειτουργούμε σαν ομάδα, όχι ο καθένας να περιορίζεται στα δικά του. Θα πρέπει μαζί να φροντίζουμε να λαμβάνονται καλές αποφάσεις, να διατηρείται το ισορροπία και να δίδεται πιο πολύ προσοχή στην κοινωνική διάσταση. Πώς μπορεί να επισέλθει τώρα αυτό στην διακυβέρνηση μέσω ανάπτυξη περαιτέρω των κοινωνικών δικτών. Θα πρέπει να φροντίσουμε και αυτό αναφέρεται στην επιστολή για την αποστολή μου. Ότι όταν διεξαγάγονται οι αναλύσεις των εξαμήνων, οι κοινωνικοί δείκτες να λαμβάνουν πιο πολύ βάρος και πιο πολύ προσοχή. Αυτό θα το κάνω από κοινού με τον συνάδελφό μου για τα οικονομικά και θα πρέπει αυτό να εκφράζεται καλύτερα στις συστάσεις χώρα. Θα πρέπει να φροντίσουμε και αυτό είναι κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να καταπολεμήσουμε την φτώχεια. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε όχι μόνο το φαινόμενο, αλλά και τα αίτια των ανισοτήτων. Και γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε ικανότητες σε ό,τι αφορά την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Όλα τα μέσα αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε και τέλος θεωρώ ότι αν ε, χρειαστεί να καταρτήσουμε ένα μακροοικονομικό πρόγραμμα ενίσχυσης για χώρες, σας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί αυτό στο μέλλον, αλλά αν χρειαστεί θα πρέπει, αυτό έχει συμφωνηθεί και αυτό θα το φροντίσουν να φροντίσουμε να υπάρχει και κοινωνική αξιολόγηση, να υπάρχει κοινωνική αξιολόγηση των μέτρων. Αυτό θα το φροντίσω προσωπικά. Και κλείνει το μικρόφωνο της ομιλητρία. Συγγνώμη, να δώσω το λόγο στην Τσιάννα Μπεκίν του EFTD. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, η Ευρώπη έχει αλυσοδεθεί από το Σύμφωνο Σταθερότητας, από το Six Pack, το Fiscal Compact και επενδύσεις για την έρευνα, την ανάπτυξη της απασχόλησης είναι προτεραιότητά σας και θα πρέπει να βγουν από το 3% του υπολογισμού των στόχων διότι είναι δαπάνες που δημιουργούν θέσεις εργασίας και πλούτο με τρόπο πολύ ανώτερο από, τον από το πρόσθετο χρέος που δημιουργούν. Θα ζητήσετε, κύριε Επίτροπε, αυτές οι επενδύσεις να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του υπερβολικού ε, χρέους και του ελλείμματος. Μια άλλη ερώτηση. Το πρόγραμμα για την εγγύηση για τους νέους είναι αποτελεσματικά ίσως στις μεσογειακές χώρες. Δεν ήταν αποτελεσματικό γιατί χρησιμοποιείται ένα μοντέλο που ήταν για τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Θα ζητήσετε διαφοροποίηση όσον αφορά τη μέθοδο εφαρμογής αυτού του μέσου, ανάλογα με κάθε χώρα εφαρμογής. Σε κάποιες χώρες η ανεργία των νέων είναι χρόνιο διαθροτικό πρόβλημα. Δεν πιστεύετε ότι χρειάζεται να προβλέπετε καλύτερος έλεγχος εφαρμογής του μέτρου αυτού που εφαρμόζεται με ευρωπαϊκούς πόρους. Διότι τελικά σε πολλές περιπτώσεις υλοποιείται μόνο στο σελίδα στο διαδίκτυο. Η κυρία Τάισαν, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας ε, τώρα. Σε ό,τι αφορά την ευελιξία στη δέσμη 6 μέτρων και σε όλες τις συμφωνίες για τον προπολογισμό. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το σημείο αυτό. Και εδώ έχουν γίνει εδώ στο Κοινοβούλιο πάρα πολλέ συζητήσει την περασμένη θητεία όταν και καταρτίστηκαν οι σχετικοί νόμοι. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία που περιλαμβάνεται στους κανόνες, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες. Η κρίση ε, προέκυψε σε μεγάλο βαθμό από υπερβολική χρέωση δημόσια και ιδιωτική. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, καταρχάς με καταπήγοντα μέτρα και με διαστατικά μέτρα στη συνέχεια, να τα βελτιώσουμε τα ζητήματα αυτά και θα πρέπει αυτή τη γραμμή να ακολουθήσουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα δημιουργώντας πιο πολύ χρέο. Αλλά υπάρχει ευελιξία στο σύμβουλο, στο σύμφωνο ευελιξία, στο σύμφωνο ε, ανάπτυξη και θα πρέπει στο μέγιστο βαθμό να αξιοποιηθεί αυτή η ευελιξία Θέλουμε λοιπόν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουμε το περιθώριο χρήση τη ευελιξία αυτή. Αυτό τι σημαίνει, να φροντίσουμε ότι υπάρχουν επενδύσει, αλλά δεν σημαίνει ότι κάποιε επενδύσει δεν μετρούν. Δηλαδή, αν υπάρχουν κάποιε ε, καλέ διστατικέ μεταρρυθμίσει, κοινωνικέ ε, μεταρρυθμίσει, και αν, για παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να πετύχουν κάποιου ενδιάμεσου στόχου, Θα καταγραφούν όλα αυτά, αλλά οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν και να γίνουν σεβαστές οι προδιαγραφές. Σε ό,τι αφορά τώρα την ευρωπαϊκή εγγύηση για την νεολαία, νομίζω ότι εδώ δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με μία ενιαία λύση για όλους. Το πρόβλημα είναι ότι τα θετικά προβλήματα που ήδη υπήρχαν πριν την κρίση διωγγώθηκαν από την κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις για τις χώρες, αλλά υπάρχει και ευελιξία στο πακέτο αυτό. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόσουν τα σωστά λειτουργικά προγράμματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το καθένα ξεχωριστά. Ντομινίκ Μαρτίν, μία γεγραμμένη. Μία γεγραμμένος. Ε, ακούω την ανεργία, την απασχόληση, το θέμα της εργασίας των νέων ηλικιωμένων, τη φτώχεια, τους ανέργους. Και είμαι καινούριο που τα ακούω όλα αυτά. Πρέπει να έχουμε νέα στρατηγική το 2020. Θέλουμε να μην εφαρμόζεται η πολιτική στα αποτελέσματα. Έχουμε πάρα πολλούς δείκτες και δεν έχουμε αρκετέ κοινωνικέ επενδύσει που δεν συμπεριλαμβάνονται στι επένδυσει εθνικέ. 20 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τι συστάσει του Διεθνού Γραφείου Εργασία. Πώ πώς θα γίνει, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Ποιο θα δημιουργήσει θέσει απασχόληση όμω, Ποιο προξενεί την ανεργία, τη μαζική, οι επιχειρήσει κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 80-90% όσον αφορά στις απασχόλησεις. Για να λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας των νέων να στηρίξουμε. Η παγκοσμιοποίηση, ο φιλελευθερισμός ανεξέλεκτος, τα δημιουργούν ε, τη μαζική ανεργία. Ο οικονομικός πατριωτισμός για να υπάρχει εσωτερική κατανάλωση και παραγωγή και ο προστατευτισμός ολογικό και φυής για την καταπολέμηση της απώλειας των τοπικών προϊόντων, της ανάπτυξης των τοπικών προϊόντων ίσως είναι η λύση. Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. Πάρα πολλά σημεία αναφέρατε. Εγώ βασικά άκουσα την τελευταία σας ερώτηση και ακούω τον πατριωτισμό και το κλείσιμο των συνόρων. Αυτή είναι η τάση που διαπιστώνω και θα ήθελα να σας παραπέμψω σε αυτά που είπα εισαγωγικά. Δεν μπορείτε να περιμένετε από εμά ότι θα σας δώσω απλοϊκές απαντήσεις, δεν θέλω να το κάνω αυτό, για σύνθετα προβλήματα. Θεωρώ ότι το πρόβλημα της ανεργίας είναι πολύ πιο σύνθετο από αυτό που κάποιες φορές παρουσιάζεται. Και αυτό έχει να κάνει με μια κοινωνία σε μεταβατική φάση με την παγκοσμιοποίηση έχει να κάνει με τις τεχνολογικές αναπτύξεις, ε, εξελίξεις, με τις εξελίξεις σε επίπεδο πληροφορικής. Όλα συμβαίνουν σε διαφορετικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να ανακόψουμε αυτή την τάση. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βρούμε απαντήσεις. Να προετοιμαστούμε και να συμμετάσχουμε. Αυτή την πρόκληση διατεθειμένη να αποδεχτώ. Να γίνουν επενδύσεις, να γίνουν προσαρμογές προκειμένου να είμαστε προσαρμοσμένοι και προετοιμασμένοι. Και με τον τρόπο λοιπόν αυτό να προετοιμάσουμε την κοινωνία μας και να διατηρήσουμε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Αυτή είναι η πρόκληση την οποία και αποδέχομαι. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ο Ζορς Μπαχ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω Μαριάν Τάισεν. Ένας από τους στόχους της στρατηγικής 2020 είναι, έχει να κάνει με την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της φτώχειας και η καταπολέμηση των επισφαλών θέσεων εργασίας. Μία ακραία μορφή τέτοιων επισφαλών θέσεων εργασίας θα μπορούσε να επιφέρει την ε, να καταλήξει σε άστεγους, πραγματικά να χάσει κάποιος το σπίτι του. Πάνω από 400.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άστεγοι. Πώς λοιπόν σκοπεύετε να βοηθήσετε τον κόσμο αυτό ο οποίος απειλείται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και δεύτερη ερώτηση. Τι θέλετε ότι μπορεί να γίνει για να διατηρηθεί η ασφάλεια και να βελτιωθεί μακροπρόθεσμα η ασφάλεια των εργαζομένων σε ευέλικτα εργασιακά περιβάλλοντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε Μπαχ. Η φτώχεια ναι, είναι όντω ένα μεγάλο πρόβλημα. Μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ήταν στόχος μας στην στρατηγική του 2020, αλλά δεν προσεγγίσαμε του στόχους μας. Μάλλον η κρίση μας απομάκρυνε από τους στόχους μας πολύ σοβαρό το θέμα αυτό και θα πρέπει να το αναλάβει ως πρόκληση η Μεροντική Επιτροπή γιατί στην πολιτισμένη κοινωνία δεν υπάρχει χώρος για τόσο μεγάλο ρυθμό ατόμων που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Ρωτάτε συγκεκριμένα για τους αστέγους. Τι μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Άτομα που δεν έχουν στέγη. Αυτοί είναι σε εξαιρετικό αποκλεισμό και χρήζουν πραγματικά έκτακτες βοήθειας. δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα το να δημιουργηθούν ε, τέτοια κέντρα, για παράδειγμα. Είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά μπορούμε να συνδράμουμε μέσω των διευθυντικών ταμείων σε ό,τι αφορά τη στέγαση, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση έργων που απευθύνονται ιδιαίτερως στους αστέγους και έργα που έχουν να κάνουν και με την ενεργειακή διαμόρφωση με καλύτερο τρόπο, για παράδειγμα, των συστημάτων στέγασης, γιατί και αυτό φυσικά παίζει ρόλο. Υπάρχουν διάφορα πειράματα λοιπόν στο επίπεδο αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να φροντίσουμε να υπάρχουν λιγότερα επισφαλή συμβόλαια εργασία. Είναι δύσκολο φυσικά αυτό σε κύριους κρίση. Σε κάποιε περιπτώσει καλύτερα να έχει κάποιο μια επισφαλή θέση εργασία και ένα επισφαλές συμβόλαιο από να μην έχει τίποτα αλλά αυτό θα πρέπει να είναι εξορισμού κάτι προσωρινό. Θα πρέπει να αποτελεί ένα βήμα προς μια πιο σταθερή κατάσταση. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε να δούμε τι γίνεται σε, κράτη, σε επίπεδο κρατών μελών. Να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα στα κρατημέλη για να καταπολεμήσουμε αυτή την τμηματοποίηση της αγοράς εργασίας. Γιατί υπάρχουν άτομα που, προσαρμόζονται, που προστατεύονται πάρα πολύ καλά στην αγορά εργασίας, αλλά υπάρχουν και άτομα που δεν μπορούν να μπουν στον τομέα αυτά της καλής προστασίας στα εργασιακά. Θα πρέπει λοιπόν σε ό,τι αφορά τις επισφαλείς ε, και κόβεται το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Ο Γκυγιόν Μπαλάς από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Κύριε Τίσεν, πριν από λίγο ακούσατε το, την εθνικιστική ρητορική μερικών και στην πατρίδα μου και πολλοί άνθρωποι εστερνίζονται πολλοί συμπολίτε μα, ιδιαίτερα όταν είναι άνεργοι βρίσκονται σε επισφαλή έθραστη κοινωνική κατάσταση. Λέμε τώρα να παροτρύνουμε τα κρατημέλη, να τα στηρίξουμε, να ευνοήσουμε την ανάπτυξη αγορά. Εμεί, οι σοσιαλιστέ και δημοκράτε, θεωρούμε ότι πρέπει να περάσουμε σε δεσμευτικέ ενέργειε. Για την εγγύηση για του νέου, για παράδειγμα. Πολλά κράτη δεν ε, προβλέπουν κατάλληλα κονδύλια για την ε, εγγύηση των νέων ή τα κονδύλια αυτά τα χορηγούν για άλλους σκοπούς. Υπάρχει μόνο στα λόγια και όχι στα έργα, δυστυχώ, αυτή η πρόβλεψη. Τι μπορεί να κάνει εμπράκτο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από το 2016 το θέμα τη πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα γίνει πιο οξύ. Τι θα προτείνετε, όχι μόνο ως ενάυσματα ή επαφιόμενοι στην ελεύθερη προαίρεση των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε δεσμευτικά μέτρα. Δεν θα πρέπει να γίνει ο τελευταίος τροχός της αμάξης η πρωτοβουλία αυτή για την εγγύηση των νέων. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Η υπόσχεση που έχουμε δώσει στους νέους για τις συστάσεις για την εγγύηση για την νεολαία είναι ασφαλώς μια πολύ σοβαρή υπόσχεση και είναι μια υπόσχεση η οποία έχει μεγάλες επιπτώσεις και όλοι θα πρέπει από κοινού να προσέξουμε ως θεσμικά όργανα, ως πολιτικοί, προκειμένου να εφαρμοστούν όλα αυτά. Να υπάρχουν αποτελέσματα αυτά προκειμένου νέοι ναι να δουν ότι υπάρχουν καρποί από την εγγύηση αυτή. Ιδάλλως θα χάσουμε μια γενιά. Θα χαθεί η εμπιστοσύνη της γενιάς αυτής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανησυχώ και εγώ γι' αυτό όπως και εσείς. Πώς θα το πετύχουμε αυτό. Διαθέσαμε μέσα και είναι καθήκον μας από την Γενική Διεύθυνση να παρακολουθήσουμε την διαδικασία αυτή, να φροντίσουμε τα μέσα αυτά να χρησιμοποιηθούν ως προβλέπεται. Δεν είναι δυνατόν να διαθέτουμε κονδύλια, να θεωρούμε ότι αυτόματα έχουμε πετύχει τους στόχους μας επειδή δώσαμε τα κονδύλια. Όχι, θα πρέπει τα κονδύλια αυτά να δαπανώνται για πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά. Να υπάρχουν στόχοι λοιπόν και να παρακολουθούμε τι γίνεται στα διάφορα κρατημέλη. Αν διαπιστώμουν ότι τα πράγματα δεν ε, πάνε καλά και ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποτελέσματα, θα πρέπει να παρεμβαίνουμε και εδώ δεν θα διστάσω να καλέσω σε τάξη τα κρατημέλη να δοθούν νέε κατευθύνσει, να βελτιωθούν τα προγράμματα και μπορούμε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους ε, βοηθήσουμε, να τους υποστηρίξουμε, γιατί τα κράτη-μέλη μπορούν να μάθουν και τα, το ένα από το άλλο. Υπάρχουν φυσικά πάντα διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά και ομοιότητες. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Γιατί επαναλαμβάνω όπως είπατε και εσείς, αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα θα περάσει μια πολύ βαθιά κρίση εμπιστοσύνη σε αυτή η νέα γενιά. Και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε σε μια τέτοια πολιτισμένη κοινωνία. Να μείνει χωρίς προοπτική μια γενιά και να μην ε, μπορεί να ξεκινήσει τη ζωή της αυτή η γενιά. Γιατί δεν υπάρχουν οι σωστές Ο κύριος Τζίσουαφ Κρασνοντέμσκι από τους μεταρρυθμιστέ συντηρητικού, σα ευχαριστώ. Μιλήσατε στην εισαγωγική σας παρουσίαση ε, για την ενίσχυση της κινητικότητας. Η κινητικότητα όμως των εργαζομένων έχει και κάποιες αρνητικές ε, συνέπειες γιατί αυτή η κινητικότητα είναι μονομερής. Από την Ανατολή προς τη Δύση, από, την, από τον Νότο προς το Βορρά, οι Πολωνοί πηγαίνουν στη Γερμανία στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν έρχονται οι Άγγλοι οι Γερμανοί στην Πολωνία για να αναζητήσουν θέσεις απασχόλησης. Και οι αρνητικές συνέπειες ε, είναι η διάλυση οικογενειών, ε, υποβάθμιση των εργασιακών συνθήκων, ε, ε, αύξηση εγκληματικότητας, ε, διαρροή εγκεφάλων, κοινωνικές εντάσεις. Τέτοιου είδους κινητικότητα οξύνει τη δημογραφική μας κρίση και δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μιλήσατε για αυτές τις αρνητικές συνέπειες, τις έχετε υπόψη σας, γιατί η κινητικότητα δεν έχει μόνο καλά, έχει και πολλά μειονεκτήματα. Και πώς θα αναχαιτήσετε αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα της κινητικότητας των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε για την ερώτησή σας. Η κινητικότητα όντως αποτελεί ένα ευαίσθητο σημείο αλλά και ένα σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει μια ενιαία αγορά στην Ευρώπη, ελεύθερη μετακίνηση, όχι μόνο προϊόντων και υπηρεσιών κεφαλαίων αλλά και ατόμων. Είναι ένας από τους πυλώνες της Ευρώπης, ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση και πάση θυσία να το υπερασπιστούμε είπατε από ανατολάς προς από νότο προς βορρά, αλλά και προς άλλες κατευθύνσεις. Κοιτώντας τις ροές, μας προκαλεί έκπληξη σε κάποιες περιπτώσεις ποιες χώρες χάνουν και ποιες χώρες υποδέχονται άτομα. Θεωρώ ότι η κινητικότητα παρέχει ευκαιρίες και ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την εργασιακή κινητικότητα. Έχουμε πάρα πολλού ανέργου στην Ευρώπη, αλλά έχουμε και πάρα πολλέ κενέ θέσει. Οι κενέ θέσει λοιπόν αυτέ και οι άνεργοι δεν ε, ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση και τα προβλήματα τα βλέπουμε σε διάφορα κράτη-μέλη. Αν λοιπόν μπορούμε να ε, επιτρέψουμε σε κάποια άτομα, σε ανέργους να φύγουν από μια χώρα και να πάνε σε κάποια άλλη όπου υπάρχουν και θέσεις και υπάρχει αυτή η βούληση από τα κράτη-μέλη, από τα άτομα αυτά, θα πρέπει να το προωθήσουμε γιατί έτσι γίνονται πιο ευτυχισμένα τα άτομα. Αυτό βοηθάει και τους ε, εργοδότες και τους ε, συναδέλφους. Επιλείται λοιπόν πρόβλημα καινών θέσεων σε μια χώρα και ένα πρόβλημα δυσαρέσκειας σε κάποιες άλλες χώρες. Και αυτό προκύπτει και από τις μελέτες και στη χώρα μου αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθολικά. Αυτοί που μετακινούνται, τα άτομα τα οποία φεύγουν, συνδράμουν στην ε, ανάπτυξη του ΑΕΠ σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι τα κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν ενδεχομένω. Θα πρέπει λοιπόν να μην κοιτάμε μόνο τα ευαίσθητα και τα αρνητικά σημεία, αλλά και τις θετικές πτυχές. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τα ευαίσθητα σημεία και θα πρέπει κυρίως να εστιαστούμε στα θέματα ενσωμάτωσης. Υπάρχουν λοιπόν μια νέα κουλτούρα στην Ευρώπη αλλά και πολλές διάφορες κουλτούρες. Πολιτισμική ποικιλομορφία θα πρέπει να ενσωματώνονται τα άτομα αυτά στις χώρες όπου καταφθάνουν και εργάζονται να νιώθουν ευπρόσδεκτα στην κοινωνία και να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία. Αυτό αφενός και αφετέρου θα πρέπει φυσικά να καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε κατάχρηση, οποιαδήποτε... Διακόπτη, Πρόεδρος. Μαρτίνα Λαμπεγιόβα από την Άλτε. Παρακαλώ, αν μπορείτε να εξοικονομήσετε κάποια δευτερόλεπτα, αν είχα την καλοσύνη. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, που είστε εδώ παρούσα και που απαντάτε τις ερωτήσεις. Μιλήσαμε εκτενώς για την ανεργία στην Ευρώπη και για την ανεργία των νέων όλος ιδιαίτερος. Έχω ιστορικό και εμπειρία από επιχειρήσεις και ανησυχώ για το πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μέσω βελτιώσεως της αντιστοιχίας δεξιοτήτων με θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου 2 εκατομμύρια έχουμε κενές θέσεις και πάνω από 5 εκατομμύρια νέους ανέργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να εργαστούν και δεν μπορούν να βρουν ταιριαστή δουλειά. Ή εργοδότες που δεν μπορούν να βρουν άτομα με τα προσόντα που απαιτούν για τις θέσεις του να καλύψουν. Για να έχουμε λοιπόν ικανούς ανθρώπους επενδύουν πολλές επιχειρήσεις στην απόκτηση προσόντων και στην απόκτηση και την αλλαγή προσόντων και θα προτιμούσαν να επενδύσουν στην εκπαίδευση σε πρώιμο στάδιο, σε πιο αρχικό στάδιο. Δεν υπάρχει κανένα συντονισμό μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων από τη μία πλευρά. Διακόπτει η πρόεδρο. Η ερώτηση. Τι προτίθεστε να κάνετε για να υπάρχει καλύτερη αντιστοιχία δεξιοτήτων με θέση απασχόληση στην Ευρώπη στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτή σίγουρα και θα πρέπει σε αυτή την πρόοδο, στην περίοδο να εστιαστούμε σε αυτό. Συμφωνώ με την ανησυχία σας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό και πολλοί κόσμος θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση, κατάρτιση. Εντάξει, αλλά ότι δεν χρειάζεται να κοιτάμε ιδιαίτερω τι ανάγκε τη αγορά εργασία. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε και τα δύο. Θα πρέπει να φροντίζουμε να υπάρχει γενική παιδεία, καλή, βασική παιδεία, να φροντίσουμε ο κόσμο να είναι σε θέση να μαθαίνει, αλλά θα πρέπει να έχει και ικανότητε, προσόντα τα οποία θα του επιτρέψουν μετά να εισέλθει στην αγορά εργασία, προκειμένου να υπάρχει σύνδεση μεταξύ τη εκπαίδευση και τη εργασία. Και φυσικά αυτό ιδιαίτερω ό,τι αφορά τι επαγγελματικέ καταρτήσει σε όλα τα επίπεδα και σε ό,τι αφορά την κατάρτιση και την εκπαίδευση των ενηλίκων, γιατί αυτό δεν, είναι, δεν έχει να κάνει μόνο με την αρχή της ζωής και της καριέρας κάποιου. Όχι, θα πρέπει να διατηρούνται και να αναπτύσσονται περαιτέρω οι ικανότητες αυτές. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ανέργους και τους μακροπρόθεσμα ανέργους. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τι ικανότητέ του, τα προσόντα τους. να μην τα χάνουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Διαπιστώσαμε ότι ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ αποφάσισε κάποια ζητήματα της εκπαίδευσης να τα μεταφέρει στην Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό το μήνυμα σε ό,τι αφορά δηλαδή τη μεταφορά τέτοιων ζητημάτων. Είναι σαφές το μήνυμα για τους ε, τομείς αυτούς και για τη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης και αγοράς εργασίας που θα πρέπει να είναι πολύ πιο στενή σίγουρα θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ Τάνια Γκονζάλες Γκουέ. Ευχαριστώ. Κυρία Τέισεν, δύο από τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 που αναφέρατε και προηγουμένως είναι ο περιορισμός της ανεργίας και η καταπολέμηση της στόχης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Λένε ότι οι πολιτικές λιτότητες που επιμένουν να μας εφαρμόζουν δίνουν αποτελέσματα. Τα στοιχεία όμως μας δείχνουν ότι επιτείνουν την ανισότητα, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στις χώρες του Νότου όπως η Ελλάδα και η Ισπανία που είχαμε μείωση της απασχόλησης από το 2007 10% και αύξηση της ανεργίας των νέων πάνω από το, που φτάνει στο 50%. Θέλετε να συνεχίσετε λοιπόν αυτές τις πολιτικές λιτότητες που τόσο μας απομακρύνουν από την υλοποίηση των στόχων της Ευρώπης 2020. Επιμείνετε στην κινητικότητα και μας την παρουσιάσετε σαν κάτι θετικό για, το, για τους επιχειρηματίες. Θεωρείτε ότι είναι μια αξιοπρεπής διέξοδος ε, για την ανεργία. Γιατί εμείς έχουμε πάνω από 2 εκατομμύρια μετανάστες ε, και η κινητικότητα έχει άλλο όνομα. Ονομάζεται αποδημία και εξορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν ληφθεί σκληρά μέτρα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Όλοι το γνωρίζουμε και το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Και το αντιλαμβάνομαι και εγώ γιατί πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα. Το ξέρουμε όλοι. Τα μέτρα ελήφθησαν. Τα μέτρα ήταν και απαραίτητα. Και ε, προέκυψε και μεγάλη αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών σε ό,τι αφορά του όρου και τι προποθέσει που τίθενται για τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει είναι κάτι φυσιολογικό, θεωρώ. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό στα πλαίσια τη αλληλεγγύη. Θα πρέπει να ξέρουμε επίση ότι σε, σε κάποιε χώρε που υπήρχαν μεγάλα προβλήματα, τα προβλήματα δεν προήλθαν μόνο από την κρίση, αλλά ουσιαστικά προσθέθηκαν στο βουνό των διαρθρωτικών προβλημάτων που ήδη υφίστανται. Και αυτά φυσικά δεν λύνονται σε μία νύχτα. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να, βελτιώσεις, οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει θα πρέπει να συνεχιστούν, να δούμε και να θέσουμε μακροπρόθεσμου στόχου, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τι βραχυπρόθεσμε επιπτώσει Και εδώ επισέρχεται ο παράγοντα του κοινωνικού, τη κοινωνική διασταση. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την πολιτική μα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει σταθερότητα. Δεν θα λύσουμε τα προβλήματα αφήνοντας κάθε έλεγχο. Θα πρέπει να φροντίσουμε αφετέρου να υπάρχει όμως και ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, να υπάρχει χρηματοπιστωτική σταθερότητα στον ιδιωτικό τομέα, στις τράπεζες, στα δημοσιονομικά, στους προπολογισμού. Και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευελιξία η οποία ενέχεται. Θα πρέπει να φροντίσουμε το ιδιωτικό κεφάλαιο να λάβει κίνητρα και θα πρέπει να συντονίσουμε τις πολιτικές μας προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη και η ανάπτυξη να μεταφραστεί σε θέσεις εργασίας γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθηθεί ο κόσμος και να μπορέσουν να ανακάμψουν τα κρατημέλη. Σας ευχαριστώ. Τέρε Ρέιντκε των Πρασίνων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Τάισεν, αγαπητή κυρία Τάισεν, εδώ είμαι. Αγαπητοί συνάδελφοι, Υπάρχουν κάποιες συστάσει κατά χώρα για τη μείωση του κόστου των συνταξιδοτικών συστημάτων. Εσείς πώς θα εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Λευκής Βίβλου για συντάξεις για να στηρίξετε τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουν την επάρκεια των συντάξεων των ηλικιωμένων ούτως ώστε να επιτρέπετε μια ζωή με αξιοπρέπεια και όχι φτώχεια. Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τις παρούσες πολιτικές που εμπεριέχουν αντιφάσεις, αυτέ που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις συντάξεις και πώς θα το θέσετε αυτό στους συναδέλφους σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις γυναίκες, πώς θα εξασφαλίσετε ότι τα μελλοντικά συνταξιδοτικά δικαιώματα των γυναικών θα ισούνται με αυτά των ανδρών, βλέποντας ότι υπάρχει διαφορά όσον αφορά τις συντάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι περίπου κατά μέσο όρο 39%. Και έχουμε και χειρότερα παραδείγματα όπως στο Λουξεμβούργο και στην Γερμανία. Σας ευχαριστώ. Τα συνταξιδοτικά συστήματα θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν και αυτό το τονίζουμε ιδιαίτερως στις ε, συστάσεις αναχώρα, στα πλαίσια του εξαμήνου και είναι σημαντικό λοιπόν αυτό. Αν θέλουμε να ζουν αξιοπρεπώς οι ηλικιωμένοι, αν θέλουμε να πληρούμε και να τιμήσουμε από πλευρά κρατών την αξίωση, τη δίκαιη αξίωση σε μια σύνταξη, σε μια αξιοπρεπή ε, σύνταξη θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι βιώσιμα τα συνταξιωτικά συστήματα και για να καταστούν βιώσιμα θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να βγαίνουν από την αγορά εργασία, να βγαίνουν στη σύνταξη οι άνθρωποι πιο αργά, να χρηματοδοτούνται καλύτερα τα, κρατη, τα συνταξιδικά συστήματα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν στο βαθμό του δυνατού όσο πιο πολλές συντάξεις σε δευτέρο πυλώνα γίνεται. Και εδώ θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη και έτσι θα φροντίσουμε την βιωσιμότητα, την αηφορία των συνταξιδευτικών συστημάτων προκειμένου και οι επερχόμενες γενιές να έχουν δικαίωμα και αξίωση σε μια αξιοπρεπή σύνταξη και οι σημερινοί νέοι θα πρέπει να ξέρουν ότι θα έχουν την εγγύηση μιας σωστής σύνταξης σε ό,τι αφορά το συνταξιδευτικό χάσμα, σε ό,τι αφορά το χάσμα μεταξύ γυναικών και ε, ανδρών. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό και αυτό δεν λύνεται μόνο με τη συνταξιδική νομοθεσία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε όλη την καριέρα της γυναίκας. Οι γυναίκες συμμετέχουν σε πολλές περιπτώσεις σε καθεστώς σημεία απασχόλησης. Επίσης ε, δεν έχουμε πετύχει το ίσο μισθό για ίση εργασία. Πληρώνονται λιγότερο οι γυναίκες και το αποτέλεσμα είναι ότι παίρνουν λιγότερες συντάξεις. Και το χάσμα που υπάρχουν μεταξύ των μισθών των ανδρών και γυναικών είναι 60% αλλά είναι διπλάσιο τουλάχιστον σε επίπεδο συντάξεων. Είναι απαράδεκτο αυτό, θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Αλλά και με άλλα μέσα, πέρα από την νομοθεσία για τις συντάξεις, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αγορά εργασίας. Να δίδονται σωστές ευκαιρίες για ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Πολ Νατάλ για το EFTD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, υπάρχει ένα ζήτημα στη Βρετανία. Μετανάστευση. Οι βολδοσκοπήσεις το δείχνουν καθημερινά. Η κινητικότητα των εργαζομένων ανοίγει την πόρτα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 450 εκατομμύρια κόσμο. Πέρσι και μόνο 250.000 άνθρωποι ήρθαν στην ε, Βρετανία για να διεκδικήσουν και επιδόματα. Οι περισσότεροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να το δούμε πιο σφαιρικά για να καταλάβουν όλοι στην αίθουσα. Είναι το μέγεθο αντιστοιχεί στον πληθυσμό του Στρασβούργου. Είναι κάτι που είναι μη βιώσιμο, αυξάνει την ανεργία και μειώνει τα ημερομίστια. Ερώτηση. Αν Βρετανική κυβέρνηση αναδιπραγματεύτηκε αναπαιδευόταν τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δίνατε στην, ε, Βρετανία τον πλήρη έλεγχο ε, των συνόρων της και τον πλήρη έλεγχο όσον αφορά τους Ευρωπαίους μετανάστες που εισέρχονται στη Βρετανία. Μία απάντηση με ένα ναι ή ένα όχι παρακαλώ. Αν θέλει κανείς να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, περιμένουμε και νομίζω ότι σωστά περιμένουμε ότι οι βασικές αρχές, οι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γίνονται σεβαστές από όλα τα κράτη-μέλη δεν κάνουμε αναδιαπραγμάτευση, αυτό θα συμβεί σε άλλο επίπεδο, αλλά η ελεύθερη διακίνηση είναι μια πολύ βασική, ε, ένας πολύ βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι ο κόσμος στην ε, ε, Ενωμένο Βασίλειο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ενιαία αγορά. αυτή η ενιαία αγορά δεν υπάρχει μόνο για τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και το κεφάλαιο, αλλά και για τους εργαζομένους. Και θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Και θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά με τίμιο τρόπο με δίκαιο τρόπο. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν αυτά να γίνονται με δίκαιο τρόπο, με τίμιο τρόπο, προκειμένου η πίεση στις τοπικές υπηρεσίες, στα τοπικά κρατημέλη και στις τοπικές αρχές να μην είναι υπερβολικά μεγάλη. Θα πρέπει να φροντίσουμε να εφαρμόζονται η νομοθεσία και θα πρέπει αυτό πάει χέρι-χέρι με την, ε, την προστασία των εργαζομένων και υπάρχει και συντονισμός των ε, ευρωπαϊκών κανονισμών για την αγορά εργασία και σε ό,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Αυτή η νομοθεσία εξελίσσεται στα κράτη-μέλη η βασική αρχή ότι ο κόσμο θα πρέπει να μπορεί να κινείται σε όλη την Ευρώπη και να απολαμβάνει κοινωνική προστασία, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διτηρήσουμε σε κάθε περίπτωση και θα πρέπει να φροντίσουμε σε ό,τι αφορά την οδηγία για τον κοινωνικό συντονισμό, μήπως υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες την χάνουν θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει κατάχρηση και αν υπάρχει κατάχρηση να την καταπολεμήσουμε. Αλλά η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων στην ενιαία αγορά και ότι η ενιαία αγορά αφορά και τους εργαζομένους και τα άτομα, αυτό είναι ένα πυλώνα στον οποίο δεν θέλω να τον απαρνηθώ. Ευχαριστώ. από το Έχετε το λόγο. Αγαπητή κυρία Τάισεν, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δέσμευσή σας για τα άτομα με αναπηρία. Έχετε δεσμευτεί ιδιαίτερως 10% περίπου του πληθυσμού, 80 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν με αναπηρία. Και παρόλα αυτά, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τα τελευταία χρόνια, δεν δίδονται παρκή μέσα. Ούτε καν 4% των κοινωνικών μέσων δεν ε, διοχετεύονται στα άτομα με αναπηρία. Συμφωνείτε, σας ικανοποιεί αυτό το, αυτή η κατάσταση. Ελπίζω πως όχι και πώς σκοπεύετε να την αλλάξετε και τι θα κάνετε για να βελτιώσετε τη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία. Γιατί πλήττονται όλος ιδιαίτερος από την κρίση. Βρίσκονται στο περιθώριο συχνά της κοινωνίας. Πώς θα προσπαθήσετε λοιπόν να αυξήσετε αυξήσετε τα μέσα που τους διατίθενται και πώς θα πετύχετε η πρόσβαση στα κτίρια να ε, μπορεί να δοθεί πιο γρήγορα για άτομα με αναπηρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, η κυρία Τάισε. Ναι, συμμερίζομαι την ανησυχία σας. Μιλάτε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ότι το 4% μόνο πηγαίνει για τους ε, ανάπηρους. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό. Αν σωστά θυμάμαι, υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο θα πρέπει να χορηγείται στα άτομα κατά του αποκλεισμού. 20%. Φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο τους αναπήρους, αλλά και άλλα άτομα. Αλλά όσοι έχουν περιορισμού και αναπηρίε έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Γιατί συχνά έχουν λιγότερε ευκαιρίε για απασχόληση και είναι πιο ευάλωτοι μέσα στην κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν ό,τι μέσα έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να τα διοχετεύσουμε και στα άτομα με αναπηρίες και το επόμενο έτη αν ε, επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπος θα το φροντίσω αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν καταρχάς. Θα πρέπει να εξετάσουμε εάν εφαρμόζονται οι συμφωνίες που έχουν ήδη αποφασιστεί και κατά πόσο υπάρχει προσβασιμότητα προκειμένου να γνωρίζει ο κόσμος τα δικαιώματά του και να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Υπάρχει το θέμα της προβασιμότητας στα κτίρια. Σίγουρα μπορούμε να μάθουμε πολλά σε επίπεδο κρατών μελών ο ένας από τον άλλον. Αλλά να υπάρχει και μεγαλύτερη προσβασιμότητα για κάποια προϊόντα σε ό,τι αφορά τους αναπήρους. Και εδώ υπάρχουν μεγάλα προσκόμματα στην ενιαία αγορά, το διαπιστώνω αυτό. Και αυτό τι σημαίνει λιγότερες καινοτομίες, πιο ακριβά προϊόντα για άτομα που τα χρειάζονται, για να είναι κινητά, να μπορούν να κινούνται για να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία. Και εδώ λοιπόν σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για την ενιαία αγορά μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα. Και σίγουρα θα σας υποστηρίξω στην τρέχουσα θητεία και το συντομότερο δυνατόν θα υποβάλω σχετική πρόταση. Ε, σας ευχαριστώ. Όλε Κρίστενσεν. Η επισφαλής απασχόληση και οι φτωχοί εργαζόμενοι επηρεάζουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο πρόεδρος Γιόγκερ ανέλαβε τη δέσμευση της, του ίσου μισθού για ίση επασχόληση στον ίδιο εργασιακό χώρο. Βέβαια δεν ήταν πολύ ε, σαφή τα σχέδιά σας. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ε, που θα αναλάβετε για να προφυλάξετε ε, τους ε, εργαζόμενους από επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, είναι ψευτοαπασχόληση, οι ε, ε, επισφαλείς συνθήκες εργασίας και πώς θα προωθήσει το θέμα της κινητικότητας σε τομείς που πλήττονται από υπερβολικά μακρά ώρα εργασίας όπως είναι το προσωπικό πτήσης. Σας ευχαριστώ σε ό,τι αφορά τις, ε, στα συμβόλαια αυτά. Ξέρω ότι είναι μια πρακτική η οποία υφίσταται σε κάποιες χώρες, σε κάποιες άλλες χώρες απαγορεύεται. Αλλά σε άλλες δεν απαγορεύεται. Νομίζω ότι πρόκειται για κάτι το οποίο αποτελεί ένα νέο φαινόμενο και πάλι θα πρέπει να το εξετάσουμε καλά, να μην κάτσουμε να το εξετάσουμε πέντε χρόνια, αλλά να το εξετάσουμε επαρκώς για να διαπιστώσουμε αν γίνονται καταχρήσεις ή όχι. Γιατί μας απασχολεί αυτό. Τα κρατημέλη μπορούν να καταρτίζουν τη σχετική νομοθεσία, αλλά έχουμε και ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία θα κράτη-μέλη μπορουν να τηρείται. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτά τα συμβόλαια μηδενικών ορών συνάδουν με κάποιους κανόνες που έχουμε κανόνες για το ωράριο εργασία, το ωράριο για τους κανόνες ε, γραπτών ε, συμβάσεων κτλ. Σε ό,τι αφορά τους ψευδοαπασχολούμενους τώρα. τώρα. Είναι σαφές. Ε, δεν σέβονται την νομοθεσία και γιατί είναι ψευδοαπασχολούμενοι, γιατί θέλουν να γλιτώσουν, να ξεφύγουν από τους κανόνες τους οποίους συμφωνήσαμε από κοινού. Που ισχύουν στα κρατημέλη για να προστατευτεί ο κόσμος, για να προστατευτεί ο εργαζόμενος από τον εργοδότη για να φροντίσουμε την ε, υγεία και την προστασία στο χώρο εργασίας, για να φροντίσουμε για το συνδυασμό του επαγγελματικού και του ιδιωτικού βίου. Είναι απάτη, θα πρέπει να, να καταπολεμηθεί. Και όχι σε κάποιου μόνο τομεί, αλλά σε όλου του τομεί. Και θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε μεταξύ κρατών μελών προ την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν πολλοί κινητοί τομεί όπου υπάρχει εργασία διασυνοριακή καταξοχή. Εδώ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο. Αλλά και πάλι θα πρέπει να συνεργαστούν οι υποπτικέ αρχέ των κρατών μελών και να φροντίσουμε οι εποπτικές υπηρεσίες των διαφόρων κρατών μελών να εμπιστεύονται πιο πολύ με μεν τους δεν. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή θα είχαμε πετύχει ένα πολύ σημαντικό βήμα για τα επόμενα χρόνια. Thank you. Σας ευχαριστώ. Μας έχουν απομείνει 20 ομιλητές. Αν περιοριστείτε στην υποβολή ερωτήσεων και όχι στην εκφώνηση λογιδρίων και αν δώσουμε και στην ε, υποψήφιο επίτροπο ΤΕΙΣ τη δυνατότητα να δώσει απλώς απαντήσεις, θα καταφέρουμε να τηρήσουμε το χρόνο. Η κυρία Γιάννα Σιτσνάσκα από, το, από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Προτινόμενη Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ήπειρος γυράσκει και μέχρι το 2016 ο πληθυσμός άνω των 60 θα είναι το 1 τρίτο του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε οι απαιτήσει ε, για της κοινωνικής πρόνοιας, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ε, θα αυξηθούν ε, δραματικά. Ε, βέβαια, σε θέματα παροχής φροντίδας ίσως δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Ποιες είναι οι ιδέες που έχετε για να στηρίξετε θέσεις απασχόλησης είτε με χρήση διαρθρωτικών ταμείων, είτε με άλλους μηχανισμούς προκειμένου να εξασφαλίσουμε ποιοτική παροχή υπηρεσιών που θα σέβονται και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κοινωνία γυράσκει και θα πρέπει να φροντίσουμε να δοθούν απαντήσεις στις ερωτήσεις και στα ερωτήματα. Αυτό φυσικά αποτελεί σε πρώτη φάση καθήκον των περιφερειών και των κρατών μελών. Δεν έχουμε αρμοδιότητα για να επεκτείνουμε αυτή την προστασία, αλλά μπορούμε να συνδράμουμε τα κράτη-μέλη και θα τα υποστηρίξουμε. Και έχουμε κάθε λόγο να το κάνουμε αυτό. Όλοι ξέρετε ότι αν η φροντίδα για τους ηλικιωμένου δεν παρέχεται σε υπηρεσίες, ο κόσμος αναγκάζεται να φροντίσει ο ίδιος ε, την οικογένειά του, τους ηλικιωμένους στην οικογένειά του και αυτό τι σημαίνει ότι δεν, δεν μπορούν να εργαστούν. Και αυτό τι σημαίνει ότι δεν λαμβάνουν οι ηλικιωμένοι το επίπεδο φροντίδας το οποίο τους αναλογεί στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία λοιπόν να καθυστερήσουμε. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα κράτη-μέλη να υποστηριχθούν για να αναπτύξουν τέτοιες υπηρεσίες. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και σε ό,τι αφορά τα αντιρρητικά ταμεία αλλά και το κοινωνικό ταμείο θα πρέπει να αξιοποιηθούν προκειμένου να δημιουργηθούν ομάδες να μαθαίνουμε ημέν από τους δε πιο πολλά προκειμένου να απτύξουμε νέες μορφές υπηρεσιών να υπάρχει και εδώ καινοτομία και όπως είπατε σωστά μπορούμε να δημιουργήσουμε και εδώ θέσεις απασχόλησης στην τεχνολογία, στις πράσινες θέσεις εργασίας αλλά σίγουρα και εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας σε ό,τι αφορά τον τομέα φροντίδας των ηλικιωμένων. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τα κρατημέλη από τα ταμεία που έχουμε και να μάθουν κυρίως το ένα από το άλλο προκειμένου γρήγορα να αναπτυχθούν και να έχουν γνώση και επίγνωση του πώς μπορούν να παρέχουν τη φροντίδα αυτή. Και μετά επαφείται στα κρατημέλη και στις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Γιάννα Τούμ από την uh, Ευχαριστώ. Η διάκριση στην απασχόληση είναι μια πρόκληση για την οικονομική απόδοση της Ένωσης και την αποτελεσματικότητά σας και στο να έχει να δημιουργεί προβλήματα στην εκπαίδευση, κατάρτιση και την ανάπτυξη. Διακριτικές πρακτικές υπονομεύουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Χρειάζεται καταπολέμηση της διάκρισης, διάκρισης σκία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φύλλο, ηλικία. Η καταπολέμηση της διάκρισης βρίσκεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Πικίλη η κατάσταση από χώρα σε χώρα όμως. Και υπάρχουν ανεπαρκές, χρειάζονται επαρκεί πολιτικέ κατά τη διάκριση εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό. Τι θα κάνετε για να εφαρμόζονται οι οδηγίες κατά της διάκρισης, τι είδου συνεργασίε θα έχετε με τον Επίτροπο για Δικαιοσύνη, καταναλωτές και Ισότητα των Φύλων για να καταπολεμηθεί η διάκριση στην απασχόληση και σε συναφείς τομεί. Ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η διακρίση είναι κάτι που απαγορεύεται στο νομικό μας σύστημα. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να μην υπάρχει περιθώριο για διάκριση. Έχουμε λοιπόν νόμοι και καταρχά θα πρέπει να φροντίσουμε να εφαρμοστούν οι νόμοι αυτοί. Θα πρέπει να κοιτάξουμε σε επίπεδο κρατών μελών κατά πόσο η νομοθεσία αυτή όχι μόνο έχει μεταφερθεί αλλά και στην πράξη εφαρμόζεται. Αν δεν συμβαίνει αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης και καθοδήγησης. Και σε αυτήν την πτυχή θα με βρείτε συμμαχό σας μαζί με τους, με τους ε, συναδέλφους της, από την Επιτροπή, με τους συναδέλφους που ήταν υπεύθυνοι για θέματα δίκαιων ευκαιριών. Η διακριτική μεταχείριση λοιπόν δεν πρέπει να έχει κανένα περιθώριο και καμία θέση στην κοινωνία μας. Μιλάμε για την ίση αντιμετώπιση των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι ε, έχουν ίδια δικαιώματα και στην στο εργασιακό πλαίσιο και θα κάνω οποιαδήποτε προσπάθεια μπορώ στα πλαίσια της Μελλοντικής Επιτροπής προς την κατεύθυνση αυτή. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νεοκλής Ηλικιώτης της ΓΚΟΕ. Σε περισσότερο από ένα σημείο το γραπτό σας απαντήσω προς την Επιτροπή να αναφέρεστε στην αντιστοιχία του εργατικού δυναμικού και των θέσεων εργασία, λέγοντα μάλιστα πως η εξάλληψή τη θα δώσει λύση στη δομική ανεργία. Τη δομική αργία κατενά οψή μα την προκαλούν οι πολιτικέ λιτότητα αλλά και η υπαγόρευση τη οικονομική πολιτική των κρατών μελών από τι Βρυξέλλε, οι οποίε δεν επιτρέπουν από κάθε κράτο μέρο να προσαρμόσει τι οικονομικέ του πολιτικέ στι δικέ του ανάγκε και δυνατότητε. Στον νότο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στι χώρε που πέρασαν ή περνούν από μνημόνια, οι μιση καταραιου τα δικαιώματα των εργαζομένων δέχονται ανελαιή επίθεση, οι εργασιακέ σχέσει απορριθμίζονται, και περιφρονείται η εργατική διαβούλευση, παραβιάζονται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων ακόμα και από τι κυβερνήσει. Αναφέρατε προηγουμένω σε απάντησή σα για την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη στον Νότο την νιώθουν οι τραπεζίτε και όχι οι εργαζόμενοι. Και το ερώτημα μου είναι πώ λοιπόν προτίθεστε να αλλάξετε την πολιτική απασχόληση τη Ένωση για να πετύχετε ασφαλή και αξιοπρεπή θέση εργασία και να διασφαλίσετε την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ιδιαίτερα στι χώρε του Νότου. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Συνάδελφε, αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι κάποια από τα κράτη-μέλη ε, υπέφεραν και επλήχθησαν ιδιαιτέρως από την κρίση και από, τα, από τις επιπτώσεις της κρίσης. Μπορούμε να το αποδώσουμε αυτό στα έκτακτα μέτρα αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε βασικά στα αίτια της κρίσης. Δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ένα από τα πράγματα που μπορώ να υποσχεθώ και θέλω να υποσχεθώ και τα οποία ζήτησε και ο Ζαν Κλοντ Juncker για να συνεργαστώ μαζί του είναι να φροντίσουμε όταν αξιολογούμε τα κράτη-μέλη να φροντίσουμε να υπάρχουν πιο πολλοί κοινωνικοί δείκτες και να, δι... να υπάρχει καλύτερη θέση και τοποθέτηση των κοινωνικών δεκτών αυτών σε ό,τι αφορά τι συστάσεις αναχώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει σε κάθε χώρα. Να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε κάθε χώρα. Και αυτό τι σημαίνει. Να μην κοιτάμε μόνο στατιστικά στοιχεία, αλλά να κάνουμε και ανάλυση εις βάθος όταν διαφέρονται κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Αυτό αφενός. Και με τη γνώση αυτή, την εις βάθος γνώση, θα πρέπει να κάνουμε καλύτερες συστάσεις και να δίνουμε καλύτερη υποστήριξη. Κάτι άλλο. Κατά δεύτερον, και αυτό σημαντικό το είπατε ότι αν θα πρέπει να υπάρξουν ε, μέτρα και προγράμματα για κρατημέλη να υπάρχει μια κοινωνική ανάλυση αντικτύπου. Ξέρουμε ότι με την Τρόικα και με τα έκτακτα μέτρα αναγκαστήκαμε να δράσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Στη μέση της θύελας λάβαμε μέτρα και πολλά σχόλια μπορούμε να κάνουμε. Όχι μόνο από εμένα. Όχι μόνο εγώ μπορώ να κάνω σχάλια. Κάναμε ολόκληρε εκθέσει εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο και ασκήθηκε κριτική σε ό,τι αφορά την νομιμότητα, τη δημοκρατική νομιμότητα και τις συνέπειες των μέτρων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν με ανοιχτό πνεύμα και χωρίς παροπίδες να τα κοιτάμε αυτά. Το χειρότερο έχει περάσει, αλλά τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί όμως ακόμα. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε με καλύτερη γνώση της κατάστασης στα κρατημέλη και με μεγαλύτερη προσοχή για την κοινωνική διάσταση, να συνεχίσουμε την ε, πολιτική μας που θα μας βάλει σε ένα βιώσιμο μονοπάτι σε ό,τι αφορά και τις θέσεις απασχόλησης. Γιατί αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα, ότι υπάρχει έλλειψη θέσεων απασχόλησης στην ε, ανάπτυξη λοιπόν στην Ευρώπη θα πρέπει να σημαίνει και επένδυση στις χώρες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα σήμερα. Η Καρή Μαντελή, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρία Τίσεν και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαι. Με βλέπετε. Πολύ ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που έχω απέναντί μου μια γυναίκα γιατί έχουμε ελάχιστες ε, γυναίκες στην Επιτροπή μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Επιτροπή μας. Η ερώτησή μου είναι ευθεία. Οι διαπραγματεύσει που γίνονται για τα ΤΤΙΠ, τη Διατλαντική Συμφωνία Τερικής Σχέση, ε, μάλλον θα θυσιάσουν τι κοινωνικέ προδιαγραφέ και ανησυχούμε γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν εγκρίνει ακόμη, δεν έχουν κυρώσει ακόμη την σύμβαση του, Διεθνή της Διεθνής και ελπίζω να το κάνουν πριν να συνάψουμε συμφωνία στα TTIP για τις επενδύσεις και το εμπόριο με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να παραλείψουμε τις κοινωνικές προδιαγραφές, ε, γιατί σε καμία ούτε εθνική νομοθεσία ούτε στην ενωσιακή νομοθεσία δεν θα πρέπει να υποβαθμίσουμε ή να απαξιώσουμε τις, ε, τους κοινωνικούς κανόνες. Σας ευχαριστώ. Διαπραγματεύσει για το TTIP, για τη συμφωνία TTIP θα πρέπει να ξαναξεκινήσουν όταν θα ξεκινήσει και να λάβετε καθήκοντα τη Νέα Επιτροπή. Η αρμοδιότητα είναι τη συναδέλφου Μάλμστρομ, όπως γνωρίζετε, αλλά και η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης ε, συμμετέχει. Δεν κοιτάμε μόνο λοιπόν θέματα εμπορίου, αλλά και κοινωνικών προτύπων. Και συμμετέχουν όσοι γνωρίζουν τα πράγματα και όσοι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Αυτό λοιπόν για να σας καθησυχάσω ότι λαμβάνεται υπόψη και αυτή η πτυχή. Κατά δεύτερον, ξέρω ότι έχει συμφωνηθεί να κινηθούμε προς μια συμφωνία, αλλά σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι δεν ε, είναι δυνατόν για να προσελκύσουμε επενδύσεις να ρίξουμε τα πρότυπά μας. Δεν είναι αυτό σκοπός μας και θα πρέπει να το συμφωνήσουμε αυτό. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε κρατός μέλος έχει το δικαίωμα νομοθεσίας στην επικράτειά του και στο κοινωνικό ε, κλάδο σε ό,τι αφορά τα βιωτικά ζητήματα. Αναφερθήκατε στα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Εδώ δεν βρισκόμαστε σε θέση άμυνα, αλλά σε επιθετική θέση. Εμείς ζητούμε από τι ΗΠΑ να κυρώσουν συμφωνίες του ΠΟΕ και να προσχωρήσουν σε αυτές. Για τη τελική ανάλυση σκοπός μας ποιος είναι αν υπάρξει συμφωνία TTIP να τονώσει τα εργασιακά πρότυπα παγκοσμίω αυτό. Και οι συνθήκες του ΠΟΕ αποτελούν ένα καλό σημείο εκκίνησης. Αυτό λοιπόν θα το προσέξουμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ανησυχούμε για τα βιωτικά μας πρότυπα, αλλά και για τα άλλα πρότυπα σε ό,τι αφορά την ποιότητα των τροφίμων. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να, ανησυχήσουμε, να ανησυχούμε για τα πρότυπα αυτά και την ενδεχόμενη επιδείνωσή τους. Ευχαριστώ, Πολ Νάταλ, του EFTD. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε πολύ ειλικρινή και λεπτομερή απάντηση στην πρώτη ερώτησή μου. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει αναδιαπραγμάτευση τη κινητικότητα των εργαζομένων και τη ελευθερία διακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχωράμε. Δύο ερωτήσει ακόμα. Υπάρχουν ιεσδήποτε παραχωρήσει που θα δίνατε στον Ηνωμένο Βασίλειο για την κινητικότητα των εργαζομένων, τόσο ώστε να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν μπορεί να δεχτεί την ελευθερία τη διακίνηση και του κανόνε και απεριόριστη κινητικότητα εργαζομένων μετά από αναδιαπραγματεύσει, Πιστεύετε προσωπικά ότι το Ηνωμένο Βασίλειο τότε θα πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφοι, αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορείτε να απευθύνετε σε μένα. Δεν μπορώ να το αποφασίσω εγώ αυτό. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε κανόνες, ότι υπάρχει συνθήκη και υπάρχει πραγματικά βασικές αρχές. Αυτές οι βασικές αρχές θα πρέπει να διατηρηθούν γιατί Ιδάλλως θα υπονομευτεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και αυτό δεν είναι σκοπός μας σε καμία περίπτωση. Αλλά ξέρω και ότι ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ είπε ότι δεν, ε, είναι, δεν κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα που έχουν κρατημέλη. Μιλάμε λοιπόν με τα κρατημέλη, κοιτάμε τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά μην περιμένετε σήμερα να σας δώσω προκαταβολικά μια απάντηση. Ξέρω ότι θα κάνω ως επίτροπος συγκεκριμένες προτάσεις. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να προτείνω να φύγει το Ενωμένο Βασίλειο. Σκοπός μας είναι να ενώσουμε τους λαούς και τις χώρες. Δεν μπορεί να είναι σκοπός μας να διώξουμε χώρες και λαούς. Άρα ας συνεχίσουμε να μιλάμε ένα τον άλλον, να ακούμε ένα τον άλλον και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αλλά σε πρώτη φάση να μιλάμε και να συζητάμε και να διαβουλευόμαστε για να βρούμε σωστές λύσεις. Ευχαριστώ. Ντανούτα Γιασλοβεύκα, τη συνάδελφα εδώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τάισεν, ε, μόλις επέστρεψα από μια διακοινοβουλευτική διάσκεψη όπου ακούσαμε από οικονομολόγους και πολιτικούς πόσο σημαντική είναι, είναι οι επενδύσεις ε, στην οικονομία και πόσο σημαντική είναι η εσωτερική κινητικότητα στην εσωτερική αγορά. Και χαίρομαι που και για σας τα σημεία αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γνωρίζουμε κυρία Τάισεν ότι για να φτιάξουμε ε, ένα ασφαλές σπίτι σημαντικά είναι τα θεμέλια του. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ασχολούμαστε με πολλά θέματα και μεταξύ άλλων ε, και με την οδηγία για τις αποσπάσεις. Τα θεμέλια της όμως δυστυχώς είναι αρκετά σαθρά. Και η οδηγία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και πολύ συχνά δεν επιτρέπουν λύσεις στο πρόβλημα. Θα πρέπει να γίνουν μελέτες και εξέταση και σε τοπικό επίπεδο για να δούμε πραγματικά την εικόνα της κατάστασης και να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις και σε τοπικό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να εμπλέξουμε και τους τοπικούς φορείς στις εργασίες, στις ε, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί οι τοπικές αυτοδιοικήσεις ε, ε, πολλές φορές δεν έχουν γνώση των σημαντικών ε, γράφων προ ανατολισμό όπως είναι η στρατηγική του 2020 και δεν ξέρουν πώς να τα εφαρμόσουν. Ευχαριστώ. Eh, Σας ευχαριστώ κύριε Γιαζοβιάσκα. Η γνώση ασφαλώς αποτελεί την καλύτερη βάση για την πολιτική. Λέτε ότι λείπουν κάποια στοιχεία, ότι δεν έχουμε επαρκείς γνώσεις. Άρα, πρώτον καθήκον μας είναι να συλλέξουμε τις γνώσεις αυτές. Για να ξέρουμε τι συζητάμε. Το είπα σε διάφορες περιστάσεις ήδη. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών. Και θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι σε βάθος η γνώση αυτή. Αυτό λοιπόν αφενός. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να συμμετέχουν οι τοπικοί φορείς. Νομίζω ήδη συμβαίνει αυτό, ιδιαίτερο ό,τι αφορά την ε, καινοτομία, τα έργα. Όλα αυτά είναι προσβάσιμα για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Νομίζω όμως ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζουν προβλήματα και ότι είναι δύσκολο από πλευράς Επιτροπής να έχουμε άμεση συνομιλία και χρηματοδότηση των τοπικών αρχών. Υπάρχουν δομές και δομές συνεργασίας. Αν διαπιστώσουμε ότι η πολιτική και ότι οι ευκαιρίες που έχουμε να μάθουμε ημένα από τους δε, να ενημερωθούμε ημένα από τους δε, να συνεργαστούμε οι ικανότητες οι οποίες υπάρχουν για αξιοποίηση πόρων δεν αξιοποιούνται επαρκώς, θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να αλλάξουν τακτική. Αλλά πάντα θα πρέπει να συνεργαστούμε μέσω κρατών μελών. Αλλά στην πράξη, ασφαλώς και θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Και όντως ακούω ότι σε τοπικό επίπεδο πολλές φορές ο κόσμος δεν ξέρει τι ισχύει σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την ε, οδηγία για τα εργασιακά. Και αυτό ασφαλώς δημιουργεί στη συνέχεια επιπλέον προβλήματα. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν πολύ καλή διάδοση των πληροφοριών και θα πρέπει να υπάρχει και μέγιστη αξιοποίηση όλων των φορέων στα έργα. Και αν αυτό δεν γίνεται επαρκώς, θα πρέπει να φροντίσουμε μέσω των κρατών μελών να το πετύχουμε και να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια και μεταφορά της νομοθεσίας μας. Δίνω το λόγο στην Βίλγια Μπλίνκεβιτσιούτε για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Τάισαν, σαν αποτέλεσμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσεως και των μέτρων λιτότητας, η φτώχεια και κυρίως η φτώχεια των παιδιών αυξάνεται ταχύτατα. Το 2011 27% όλων των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινδύνευαν με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επί του παρόντος δεν αποδίδει στα μέτρα για τους πλέον ευαλότους της κοινωνίας. Ερώτηση. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα προτείνετε ούτω ώστε η Ευρώπη να μπορεί να πετύχει τους στόχους για τη φτώχεια που καθορίζονται στη στρατηγική του 2020. Ποια είναι η θέση σας όσον αφορά τη εισαγωγή εγγυήσεων για τα παιδιά, παρόμοια με το σύστημα εγγυήσεων για τους νέους, ούτω ώστε κανένα παιδί να μην μένει πίσω. Να το εξασφαλίσουμε αυτό. Ε, Σα ευχαριστώ. Τα παιδιά είναι ένα πάρα πολύ πολύτιμο αγαθό στην κοινωνία μας και αν είναι φτωχά τα παιδιά ξεκινούν άσχημα τη ζωή της και αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Και εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι η φτώχεια είναι ένα θέμα το οποίο σε μεγάλο βαθμό εμπίπτει στον τομέα αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα πρέπει να του υποστηρίξουμε λοιπόν. Το κάνουμε. Υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη μέσω συνεργασία ε, με οργανώσει για του φτωχού, μέσω των συστάσεων αναχώρα όπου λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά το πρόβλημα αυτό, όπου υπάρχει ένδια, όπου υπάρχει φτώχεια και διαπιστώνουμε ότι δεν γίνονται αρκετά. Ζητούμε μεταρρυθμίσει από τα κράτη-μέλη. Και αυτό ασφαλώς θα πρέπει να το συνεχίσουμε ακόμα πιο εντατικά στο μέλλον. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι δεν θα μας βοηθήσει μόνο η πολιτική για, τους, για τη φτώχεια. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τη γενικότερη οργάνωση της κοινωνίας, να φροντίσουμε τα παιδιά και πριν ακόμα την γέννησή τους να έχουν φροντίδα, να υπάρχει φύλαξη για τα παιδιά, να υπάρχει καλή εκπαίδευση, να υπάρχει οικογενειακή υποστήριξη και σχετικές υπηρεσίες προκειμένου ακόμα και αν η οικογένεια βρίσκεται προσωρινά σε καταστάσεις ένδυας, να υπάρχει δυνατότητα να φροντίσει τα παιδιά της. Και να μπορούν οι νέοι να έχουν μια καλύτερη προοπτική και να μην τους αφήνουμε στην τύχη τους. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε, να αναπτύξουμε καινοτόμα εργαλεία, έχουμε δυνατότητες δράσης, έχουμε και προγράμματα και σχετικά μέσα και τονίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σε ό,τι αφορά και τους στόχους του 2020 περιλαμβάνεται η φτώχεια και θα πρέπει να συνεχίσει να περιλαμβάνεται. Θα πρέπει να συνεχίσει να περιλαμβάνεται ιδιαίτερως και σε συστάσεις ανά χώρα. ευχαριστώ. από τους ε, μεταρρυθμιστές συντηρητικούς. Αξιότιμη υποψήφια επιτροπέ. Είμαστε από την ίδια μικρή περιφέρεια και αντιλαμβανόμαστε και οι δύο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι αντιμέτωπες και αντιμέτωπα με τεράστιες προκλήσεις. Παρά τη δύσκολη χρηματοοικονομική κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξεκινήσουν κάποια μεγάλα ε, έργα υποδομών για να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα κινητικότητας. Αυτό θα ωφελήσει και την οικονομία. Ποιες είναι οι δυνατότητες λοιπόν που έχει μια μικρή περιφέρεια, όπως η Φλάνδρα για παράδειγμα, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο να κάνει μεγαλόπνοες και μεγάλες κλίμακας επενδύσεις και να διανύμει το κόστος των επενδύσεων αυτών σε πολιτές επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Στέβενς, λέει η κυρία Τέισεν. Από την ερώτησή σας για... Καταλαβαίνω νομίζω, νομίζω για ποιες υποδομές μιλάτε. Ίσως ε, ο κόσμος που δεν είναι από τη χώρα που είμαστε εγώ και η κυρία Στέβενς ε, δεν καταλαβαίνει ακριβώς ποια εργανοούμε σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις που θα πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα. Νομίζω ότι εδώ το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες. Δεν μπορούμε για μια μικρή χώρα όπως το Βέλγιο ή για μια μικρή περιφέρεια όπως η Φλάνδρα να κάνουμε εξαιρέσεις και κανείς δεν νομίζω δεν θα περιμένει από μένα να αλλάξω τους κανόνες και θα ήθελα επίσης να υποδείξω ότι σε ό,τι αφορά τις δημόσιες δαπάνες και την κατάταξή τους στα δημοσιονομικά υπάρχουν πρότυπα τα οποία ελέγχονται και από την Eurostat, από μια ανεξάρτητη οργάνωση. Υπάρχουν λοιπόν κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμοστούν στη Φλάνδρα, στο Βέλγιο, αλλά όπως και στις άλλες χώρες. Η Eurostat ε, θα εξετάσει τους φακέλους και θα κρίνει με ανεξάρτητο πνεύμα, όπως κάνει και παντού αλλού. Να τονίσω και να προσθέσω, συνάδελφε, ότι ως Βελγίδα Επίτροπος θα αντιμετωπίσω ασφαλώς τέτοια προβλήματα, αλλά υπάρχουν τέτοια προβλήματα και σε άλλες χώρες. Αλλά δεν πρόκειται να αποδεχτώ εντολές από τη χώρα μου και όλα τα θέματα, άλλους τους φακέλους θα τα αντιμετωπίσω με ίσο τρόπο. Και θα ήθελα να τονίσω τη λειτουργική ανεξαρτησία της Eurostat, την οποία θα τη σεβαστώ απολύτως. Αυτό δεν είναι μόνο καθήκον μου, αλλά και πρόθεσή μου. From the Group. Ο Ιβο Βάιγκλ από τους Φιλελεύθερους. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Τίσεν. Η σημερινή ημέρα είναι η, η ημέρα των ηλικιωμένων και στο θέμα αυτό αναφέρεται και η ερώτησή μου. Θα δώσετε μάχη και θα υποβάλλετε πρωτοβουλίες προκειμένου να υιοθετήσουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική προσαρμογή στις δημογραφικές αλλαγές. Γιατί χρειαζόμαστε πολλά νέα μέσα για να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Λυπούμε που δεν έχουμε χρόνο για μια πιο ενδελεχή ανάλυση και σίγουρα οι ηλικιωμένοι δεν έχουν λόμπι και ομάδες πίεσης για να προωθήσουν τα συμφέροντά, τα συμφέροντά τους, οπότε όλα εξαρτώνται από την δική μας καλή θέληση και την καλή θέληση των κρατών μελών. Θα πρέπει να βοηθήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ καλές δράσεις. Σας ευχαριστώ συνάδελφε αναφέρεται ότι οι ηλικιωμένοι δεν έχουν αρκετά, αρκετούς οδούς, αρκετές οδούς άσκησης πίεσης. Λόμπι. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι, σε, κάποιοι στην κοινωνία έχουν τις, σωστούς, τις σωστές διόδους ε, άσκησης ε, πίεσης ε, και άλλοι δεν έχουν αυτά, δεν έχουν την ιδιότητα για να προσλαμβάνουν λομπιίστες. Θα πρέπει λοιπόν και είναι καθήκον όλων των ε, πολιτικών να ακούμε όλους τους ανθρώπους και τους λομπιίστες, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι και κάποιοι δεν εκπροσωπούνται από λομπιίστες και τα δικά τους συμφέροντα επίσης θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη και θεωρώ ότι οι ηλικιωμένοι έχουν πολλές ε, δυνάμεις, οργανώνονται πάρα πολύ καλά για να πρόσπισουν τα συμφέροντά τους και αυτό το χαιρετίζω θα πρέπει να φροντίσουμε οι ηλικιωμένοι να μπορούν να συνεχίσουν να είναι ενεργοί. Αν θέλουμε, αν περιμένουμε, αν δώσουμε δυνατότητα στους ηλικιωμένους να συνεχίσουν να απασχολούνται πιο πολύ και για τα συνταξιδικά συστήματα, προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν τις σωστές ικανότητες και τις απαραίτητες ε, προσόντα, να υπάρχει διαβίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων. Θα πρέπει να φροντίσουμε πέρα από την προθυμία τους να υπάρχουν και λειτουργικές θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους αυτούς. Θα πρέπει να γίνουν λοιπόν ε, τροποποίησεις ε, και από πλευρά των επιχειρήσεων για να επιτρέπουν στα άτομα τα ηλικιωμένα να μένουν πιο πολύ στην αγορά εργασίας. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό για να είναι ενεργός η γύρανση. Με αποδεκτό τρόπο να μένουν στην αγορά εργασία. και επίσης να φροντίσουμε για τη βιωσιμότητα των συνταξιδοτικών συστημάτων. Αλλά αυτό το συζητήσαμε ήδη και τονίζω ιδιαίτερα τη σημασία της βιωσιμότητας αυτής. E Ο Σβέν από το ΕΛΚ. Κυρία Τάισεν, και με τη δική μου ερώτηση θα έχετε την ευκαιρία να αναφερθείτε στο σημαντικό θέμα της δημογραφίας, γιατί νομίζω ότι δύο λεπτά για χρόνο απάντησης δεν φτάνει ως χρόνος. Η δημογραφική αλλαγή, όπως αναφέρατε, είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της εποχής μας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπατε, είναι αντιμέτωπη με διάφορες προκλήσεις και βλέπουμε πώς γυράσκει ο πληθυσμό, αλλά παράλληλα πώς μειώνονται και οι γεννήσεις σε πολλές χώρες οι παράγοντες αυτές έχουν διαφορετική σημασία για την κοινωνική οικονομία της αγοράς και για τα κοινωνικά μας συστήματα σε όλες τις χώρες και για την ε, πολιτική απασχόληση. Θα μπορούσατε παρακαλώ να μας ε, αναφέρετε κάποια συγκεκριμένα μέτρα για το πώς εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη δημογραφική αλλαγή σκοπεύετε να εργαστείτε. Και άλλη μια ερώτηση, επιτρέψτε μου. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο συνταξιβετικό σύστημα και πότε και διακόπτει η Πρόεδρος. Μάλιστα, να απαντήσετε κυρία Τέισεν. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε στην Ευρώπη για καινοτομία να μην σκεπτόμαστε μόνο την έρευνα, την ανάπτυξη για τη βιομηχανία. Να έχουμε υπόψη μας και την έρευνα και την ανάπτυξη για νέες υπηρεσίες, για νέες ε, μορφές πολιτικής για νέα αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Η δημογραφική αλλαγή δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα καινούριο. Το γνωρίζουμε εδώ και καιρό. Διαπιστώνουμε εκ παραλλήλου ότι σε πολλές χώρες, όχι παντού, αλλά σε πολλές χώρες ήταν πολύ καθυστερημένη η αντίδραση σε αυτό το φαινόμενο. Θα πρέπει λοιπόν να καταστεί μια προτεραιότητα αυτή σε ό,τι αφορά την κοινωνική καινοτομία. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες μορφές ανταπόκρισης. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις δημογραφικές τάσει. Υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από τα χέρια μας και τα κρατημέλη, προκειμένου να φροντίσουμε να υπάρχουν νέες κοινωνικές υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά την ε, φροντίδα και όλες τις υπηρεσίες να γίνει ένας προσανατολισμός σε όλη την κοινωνία στις δημογραφικές αλλαγές. Να φροντίσουμε να γνωρίσουμε πιο πολύ εις βάθος το φαινόμενο, να αναζητήσουμε νέες μεθόδους, να φροντίσουμε οι παράγοντες και οι εμπλεκόμενοι φορείς να είναι ενημερωμένοι, τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία μπορούμε να διαθέσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε, να υπάρξουν νέες μέθοδοι φροντίδας. Είναι πάρα πολύ ευρύ το φάσμα των δράσεων που πρέπει να λάβουμε. Δεν μπορούμε τόσο πολλά να κάνουμε σε επίπεδο νομοθεσίας, αλλά σε επίπεδο συστάσεων, σε επίπεδο ταμείων για κοινωνική κοινοτομία και κυρίως σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή βέλτιση των πρακτικών. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα κινητοποιήσουμε. Ευχαριστώ, η Πέτρα Κάμερβετ. Από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, μέλος επιτροπή Επιτροπής Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Τάισεν. Ξέρουμε ότι η υψηλή ενέργεια των νέων αποτελεί ένα καυτό πρόβλημα σε πολλά κράτη-μέλη και ξέρουμε ότι το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί με κανένα δυο ωραία προγράμματα. Χρειάζονται σωστές δομές. Και βλέπουμε σε πολλά κράτη-μέλη ότι η δυτή αυτή εκπαίδευση, δηλαδή η συνδυασμός εκπαίδευση στα σχολεία και κατάρτιση στις επιχειρήσεις έχει αποδεχτεί ανθεκτική στην κρίση Ίσως λοιπόν αυτή να είναι μία απάντηση. Προκειμένου να υπάρχει σωστή εκπαίδευση και ανάπτυξη. Ποιε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε για την προώθηση ενό τέτοιου συστήματο εκπαίδευση έχετε σχεδιάσει και πώ θέλετε να υποστηρίξετε τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν τέτοια συστήματα εκπαίδευση και ποιοι μηχανισμοί συνεργασία μεταξύ τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση και τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση θέλετε να δημιουργηθούν προ την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνουμε ότι αυτή η μορφή δυτής εκπαίδευσης μπορεί να έχει πολύ καλούς καρπούς. Ξέρουμε και από την πράξη αλλά και από την θεωρία ότι ο κόσμος αυτός βρίσκει πολύ πιο εύκολα δουλειά. Και αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων, σε ό,τι αφορά τη μετάβαση προς την αγορά εργασίας. Σίγουρα λοιπόν μπορούμε να δούμε μια λύση για το μέλλον. Τι μπορούμε να κάνουμε από πλευρά Ευρώπη. Ξέρετε ότι είναι το μέσα αρμοδιότητα των κριτών μέλων, αλλά μπορούμε να του ε, βοηθήσουμε. Με ρωτάτε συγκεκριμένα τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε ήδη συμφωνίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για διαβούλευση, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ό,τι αφορά θέματα κατάρτισης. Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για θέσεις μαθητείας. Υπάρχουν λοιπόν ήδη δρομολογημένες δράσεις, αλλά μπορούμε και περαιτέρω να συνεχίσουμε τη συνεργασία, όπως είπατε κι εσείς, με πολιτισμικούς παράγοντες. Στις επιστολές για την αποστολή μας από τον Jean-Claude θα δείτε ότι η επαγγελματική κατάρτιση και η εκπαίδευση και η διαβίου εκμάθηση και η εκπαίδευση των ενηλίκων έχει μεταφερθεί πλέον στο πεδίο αρμοδιότητας τη Γενικής διεθνής Απασχόλησης. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Ξέρουμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πρόγραμμα Erasmus Plus σε ό,τι αφορά τις ασκήσεις, τη συνεργασία, τη συνοριακή για την διοργάνωση μαθημάτων ή για τη συμμετοχή σε τέτοια μαθήματα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά τέτοια προγράμματα. Η χρηματοδότηση λοιπόν και η διοικητική εποπτεία και κλείνει το μικρόφωνο του Thank Ευχαριστώ πολύ. Ρενάτε Βέμπερ, του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επιτροπέ, εκτίμησα ιδιαίτερα την, ε, τα σχόλιά σας για την ελεύθερη κίνηση του κόσμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά την κινητικότητα την εργασιακή. Επίσης, συμφωνώ μαζί σας ότι Χρειαζόμαστε άλλου είδους εκπαιδεύσεις και επαγγελματικέ καταρτήσεις προκειμένου να έχουμε μια αντιστοιχεία της, των δεξιότητων και των αναγκών της οικονομίας. Πόσο φιλόδοξοι θα είστε και πόσο μακριά θα πάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πιέσει τα κράτη-μέλη να, να, να αλλάξουν τα προγράμματα σπουδών ή το περιεχόμενο ε, των προγραμμάτων διαβίου κατάρτισης ή εκπαίδευσης. Ε, τι μέτρα ε, σκέφτεστε να υιοθετήσετε σχετικά. Ehm, Σα ευχαριστώ κυρία Βέμπερ. Οι υποχρεώσει είναι κάτι δύσκολο. Δεν νομίζω ότι έχουμε αρμοδιότητα σε επίπεδο εκπαίδευση να αποφασίσουμε για του μαθησιακού κύκλου. για τα προγράμματα εκμάθησης, αλλά μπορούμε να υποστηρίξουμε, να παρατρύνουμε, να συλλέξουμε στοιχεία και δεδομένα και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε στο μέγιστο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και τεχνικής κατάρτισης. Τι μπορούμε να προσφέρουμε. Κυρίως ε, συλλογή στοιχείων και γνώσης σε διάφορα κράτη-μέλη. και να φροντίσουμε η γνώση αυτή να χρησιμοποιείται και σε άλλα κράτη-μέλη τα άτομα τα οποία καταρτίζουν τους, ε, τα μαθησιακά τα προγράμματα εκπαίδευση να μπορούν να μαθαίνουν οι μεν από τους δε. Και έχει φανεί στο παρελθόν ότι αυτό είναι μια πολύ καλή μέθοδος. Φαίνεται λίγο σόφτος μέθοδος, λίγο ήπια. Έτσι έχει η κατανομή των αρμοδιοτήτων. Δικαιώς μας καθήκον είναι να φροντίσουμε να υπάρχει υποστήριξη και να υπάρχει ανταλλαγή γνώσης. Να συλλέξουμε στοιχεία Πού αλλού μπορούμε να βοηθήσουμε? Στην αναγνώριση των αποτελεσμάτων, των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Έχουμε αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσφορών για τα άτομα, τα οποία ακολουθούν ένα επάγγελμα. Υπάρχει και ένα πλαίσιο, όπου υπάρχει, γίνεται μια απόπειρα ταξινόμηση ε, των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, των διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων και σχετικής αξιολόγησης. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η προσπάθεια, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να συνεχιστεί και να βελτιωθεί. Να φροντίσουμε να υπάρχει χώρος για όσα άτομα προερχόνται και από την επαγγελματική κατάρτιση, από άτυπη κατάρτιση ενδεχομένως, να μπορούμε να τα αξιολογήσουμε και να τα εκτιμήσουμε πιο σωστά τα άτομα αυτά. Και αυτό θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει για να υπάρχει αυτή η καλύτερη σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας σε συνδυασμό με την κινητικότητα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η Ράτσα Γκαρσία Πέρες για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Επιτροπή Γυναικών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Τάισερ, η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και ισότητα των φύλων είναι αναπόσπαστα στοιχεία των ε, ευρωπαϊκών πολιτικών και ιδιαίτερα της πολιτικής που αποτελεί το χαρτοφυλακίου σα. Έχουμε 16% μισθολογικό χάσμα, 39% χαμηλότερες ε, συντάξεις για τις γυναίκες από ό,τι στους άντρες και 27% των γυναικών απειλούνται με κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας. Στο κοινωνικό αυτό το οποίο θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα για να μειωθεί αυτό το τριπλό χάσμα, το μισθολογικό, το συνταξιδοτικό και το χάσμα σε ό,τι αφορά τη φτώχεια τι νομοθετικά μέτρα πρόκειται να θεσπίσετε και τι πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για να μειωθεί αυτό το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών Επίσης, πώς θα αναμίξετε, πώς θα εμπλέξετε τους άνδρες, ιδιαίτερα τους ε, συναδέρφους σας επιτρόπους, σε, αυτήν την, ε, σε αυτό το σημαντικό καθήκον εξασφάλισης της ισότητας των δύο φύλων. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, να ξεκινήσω από το τέλος. Ε, οι γυναίκες και οι άνδρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλοι θα πρέπει να φροντίσουν για ίση αντιμετώπιση και ίση μεταχείριση των ανδρών και των γενικών στην Ευρώπη. Είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο αυτό στην Ευρώπη και σε ό,τι αφορά την πρώτη πρώτη ε, συνθήκη της Ρώμης στο άρθρο 119, νομίζω το ξέρω απ' έξω, ε, είναι, τι προβλέπετε, ίσως μισθός για ίση εργασία. Βάσει αυτού του άρθρου λοιπόν αναπτύξαμε την κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Μπορούμε να καταρτήσουμε νομοθεσία και να τα προαγάγουμε όλα αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και να κάνουμε συστάσεις και θα πρέπει να τηρήσουμε τις συμφωνίες. Έχουμε πει ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι πιο διαφανείς σε ό,τι αφορά τους μισθούς γυναικών και ανδρών. Και έτσι να παρατρύνουμε την μεγαλύτερη ισότητα. Θα πρέπει λοιπόν να τα παρατρύνουμε αυτά. Τώρα κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει νομοθεσία, ήδη υπάρχει νομοθεσία. Θα πρέπει απλά να εφαρμοστεί καλύτερα, με πιο ευφυή τρόπο. Ίση εργασία για... Ίσως μισθός για ίση εργασία αυτό είναι αυτονόητο. Ακριβώ την ίδια δουλειά κάνουμε, ακριβώ τον ίδιο μισθό πρέπει να παίρνουμε. Έχει να κάνει αυτό με την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Και προ αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Οι γυναίκε συμμετέχουν λιγότερο. Απασχολούνται σε καθεστώ μη απασχόληση πιο συχνά. Επειδή θέλουν ή πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά ή άλλα άτομα στην οικογένεια. Σταματούν πιο γρήγορα τη δουλειά. Και εδώ υπάρχει διακριτική μεταχείριση σε ό,τι αφορά το όριο συνταξιοδότηση. Ε, διαπίστωσα με μεγάλη μου έκπληξη ότι έχουν ε, λιγότερα δικαιώματα σε ό,τι αφορά το όριο το οποίο μπορούν να συλλέξουν συνταξιδοτικά δικαιώματα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν ένα πιο σωστό πλαίσιο για να συμμετέχουν πιο καλά οι γυναίκε, για να μπορούν να συμμετέχουν. Να υπάρχει φύλαξη για τα παιδιά, να υπάρχουν υπηρεσίε φροντίδα ε, τη οικογένεια και άλλοι μηχανισμοί οι οποίοι εμέσως αποτρέπουν τις γυναίκες από το να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν ε, για να το πετύχουμε αυτό να συζητήσουμε πολύ ημέν με τους δε και κλείνει το μικρόφωνο της Thank you. Ευχαριστώ. Κωνσταντς Λεγκρίπ. Εκπροσωπεί το ΕΛΚ στην Επιτροπή Γυναικών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, άκουσα με μεγάλη ικανοποίηση την απάντησή σας στο ερώτημα που έθεσε η προλαλή σας. Και άκουσα και τη βούλησή σας για περισσότερη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ενώσεως. Και όσον αφορά τη διαφορά των αμοιβών, το μεγάλο, μεγάλη διαφορά μεταξύ των φίλων και για τις συντάξεις και άλλα σκάνδαλα τέτοια. Λαμβάνουμε υπόψη την βούληση που εκφράσατε. Σας ζητάμε ενδεχομένως να συνεχίσετε την απάντησή σας όσον αφορά τις βασικές ανησυχίες που υπάρχουν για τις Ευρωπαίες γυναίκες. Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα μπορούσατε να θεωρήσετε ότι μπορείτε να δρομολογήσετε μαζί με τον συνάδελφο για την ισότητα των φύλων. Ούτε ώστε να δώσετε κίνητρα στα κράτη-μέλη πρώτη να εφαρμόσουν τις ε, υφιστάμενε νομοθεσίες. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Πολύ συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι κυρίως να κοιτάξουμε τι γίνεται στην πραγματικότητα, στην πράξη επιτόπου. Νομίζω ότι αυτό που λείπει είναι η επίγνωση του τι ακριβώς συμβαίνει στα κρατη Και όποτε βλέπουμε ότι τα κρατη δεν σέβονται τους κανόνες, ότι η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται επαρκώς, ότι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου να οδηγηθούν προς μια διαφορετική κατεύθυνση συμπεριφορά στα κρατη και να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέτρο έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό λοιπόν αφενός. Καμία διακριτική μεταχείριση βάσει του φύλου. Να πω σε σχέση και με την προηγούμενη ομιλήτρια που ανέφερε την Επιτροπή. Χάρηκα όταν μου ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιούγκερ ότι ήθελε να έχει αρκετές γυναίκες στην Επιτροπή και παραπάνω από εννέα, εάν περνούσε από το χέρι του, όχι μόνο επειδή το ζητάει το Κοινοβούλιο, αλλά επειδή και ο ίδιος είναι πεπισμένος για τη σημασία αυτή ζούμε στον 21ο αιώνα και θα πρέπει να φροντίσουμε οι γυναίκες να ε, παίζουν το ρόλο τους και δεν ε, με ικανοποιεί το να υπάρχει μόνο ο ελάχιστος αριθμός γυναικών. Και η Επιτροπή λοιπόν είναι απόλυτα πεπισμένη γι' αυτό και σίγουρα θα μας υποστηρίξει και η υπόλοιπη Επιτροπή. Και μαζί με τον συνάδελφο που είναι αρμόδιος για θέματα ισότητας ε, φύλων θα φροντίσω προκειμένου όλα αυτά να επισέλθουν και στον τομέα τον εργασιακό και αν αναζητήσει σύμμαχο στο πρόσωπό μου σίγουρα θα έχει ένα σύμμαχο. Αν με, ρωτάει, αν με ρωτήσει κανείς αν είμαι φεμινίστρια, απαντάω αντιαφασβητήτα με ένα ηχηρό ναι. Ότι οι γυναίκες δηλαδή που χρειάζονται υποστηρίξη θα τη βρουν από εμάς. Νομίζω ότι είναι καθήκον μας αυτό και σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι και δική μου αποστολή. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην Έλενα Τζεντήλε από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ χαιρετίζω την αξιότιμη την κυρία Τίσεν υποψήφια επίτροπο. Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας σίγουρα είχαν συνέπειες καταστροφικές. Η ανεργία αυξήθηκε πολύ γρήγορα, οι κοινωνικές υπηρεσίες διαλύθηκαν στην πράξη με τον άκρος οδυνηρό, άκρος οδυνηρές περικοπές των κοινωνικών ωφελημάτων. Είναι απαράδεκτη κατάσταση, θα πρέπει να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε τα δίχτυα κοινωνικής προστασίας. Τα προγράμματα δημόσιας στήριξης, κανείς να μην μένει πίσω. Λοιπόν, θα δεσμευτείτε κυρία Τίσεν να θεσπίσετε ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που θα μπορεί αυτό το πλαίσιο να υλοποιήσει ένα κάποιο είδος κοινωνικού σχέδιο προστασίας που θα εγγυάται την καθολική προστασία στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες. Ένα νομικό πλαίσιο ευρωπαϊκό για τους ελάχιστους μισθούς, ούτω ώστε να είναι αξιοπρεπείς οι αμοιβέ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνετε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πολύ σημαντική αυτή ερώτηση για το κατά πόσον θέλω να ταχθώ υπέρ ενός καλού κοινωνικού πλαισίου. Ναι, υπάρχει η συνθήκη που είναι και η κατευθυντήρια γραμμή. Υπάρχει και το πρόγραμμα του Προέδρου Γιούγκερ βάσει του οποίου εκλέχθη στο Κοινοβούλιο και από τα δύο προκύπτει ότι χρειάζεται ένα καλό κοινωνικό πλαίσιο, ότι θα πρέπει να δοθεί μια σωστή διάσταση στην κοινωνική οικονομία αγοράς. Ναι, αγορά, προσφορά και ζήτηση, σύμφωνη, αλλά και κοινωνική διάσταση και μάλιστα με διαμόρφωση βιώσιμη. Αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστικότητα για δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξη. Αυτό είναι το καθήκον μας. Τώρα, το κατά πόσον θα υπάρξει ένα ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να τηρούν τα κρατημέλη, νομίζω ότι δεν μπορούμε αυτό να το διαμορφώσουμε ως ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, όλοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπει η συνθήκη σε θέματα εργασιακού δικαίου, να κάνουμε κάποιες ελάχιστες συμφωνίες σε ό,τι αφορά τα συστήματα προστασίας, προκειμένου να υπάρχει βιωσιμότητα. Όλα αυτά τα μέσα λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιηθούν και σίγουρα θα είμαστε σύμμαχοι στη διαδικασία αυτή. Μιλήσατε και για τον ελάχιστο, τον κατά το μισθό. Δεν το συζητήσαμε δεν μιλήσαμε για θέματα ελάχιστου μισθού, μιλήσαμε για θέματα ελάχιστου εισοδήματο. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε χώρα κατώτατο μισθό. Αυτό πιστεύει και ο κύριος Γιούγκερ το είχε επαναλάβει δημόσια σε διάφορες περιστάσεις. Αλλά έχουμε και το άρθρο 143.5 τη συνθήκη αν δεν κάνω λάθο, που ορίζει ότι δεν είμαστε εμεί αρμόδιοι για θέματα καθορισμού των ε, μισθών. Αλλά μπορούμε να παροτρύνουμε τα κρατημέλη γιατί ξέρουμε ότι ο κατώτατος μισθός μπορεί να αποτελέσει ένα παράγοντα σε ό,τι αφορά τον δίκαιο ανταγωνισμό ή τον άδικο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να παροτρύνουμε τους ε, κοινωνικούς εταίρους να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους για να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε οτιδήποτε σε όποια κράτη δεν έχουν τέτοιους κατώτατους μισθούς. Σας ευχαριστώ. Η Μαρία Ρένα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κυρία Τέισεν. Από την κρίση του 2008 και με ένα κοινωνικό, φορολογικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ που γίνεται τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε 16.000 αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και ε, χιλιάδες εργαζόμενους που πέρασαν στην ανεργία. Πώς θα βοηθήσουμε τα θύματα αυτών των αναδιαρθρώσεων. Κάποια κρατημέλη με τους κοινωνικούς εταίρους ε, προσπάθησαν να ενημερώσουν ε, τους εργαζόμενους ε, όπως έκανε το Βέλγιο με την νομοθεσία Ρενό. Είχαμε μάλιστα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μια νομοθετική πράξη για τη διαβούλευση και την ενημέρωση των ε, εργαζομένων εν ώψη μιας αναδιάρθρωσης. Θα προτείνεται μια οδηγία πλαίσιο εισακούγοντας το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για να προστατεύσουμε καλύτερα τη βιομηχανία μας απέναντι στον αθέμητο διεθνή ανταγωνισμό, γιατί μας μην ξεχνάμε ότι η βιομηχανία μας δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Yeah, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή που μου θέσατε. Η αναδιάτρωση αποτελεί ένα γεγονός. Πολλά έχουμε ήδη κάνει και σίγουρα πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Το πιο έξυπνο που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις. Ξέρουμε ότι κάποιες καταστάσεις θα προκύψουν. Θα πρέπει λοιπόν σε μακροοικονομικό αλλά και μικροοικονομικό επίπεδο να δείξουμε προληπτική διάθεση. Θα πρέπει να γίνουν και πιο πολλά πέρα από διαβουλεύσεις και ενημερώσεις, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να προχωρήσουν σε ενδεχόμενες αναδιαρθρώσεις και όσοι ε, ενδεχομένως χάσουν, υπάρχει, για όσους υπάρχει κίνδυνος να χάσουν τη δουλειά τους, να περάσουν από μια επανεκπαίδευση. Να δούμε τι μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο κράτους μέλους για να γίνει μια τέτοια αναδιάθρωση και το τι θα σημαίνει και για τις κοινωνικές ε, διαστάσεις, για τον κοινωνικό αντίκτυπο αυτό. Άρα, η ενημέρωση και πρόληψη. Ξέρω ότι στην έκθεση ΣΕΡΚΑΣ είχε ζητηθεί να προκύψει σχετική νομοθεσία και ξέρω ότι αυτό είναι αντίθετο. Ότι αντίθετο τελικά αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην υποβληθεί πρόταση νομοθεσία, αλλά ε, να δημορφωθεί ένα πλαίσιο. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση της εργασίας μας στην παρούσα φάση, προκειμένου να υπάρξει αυτή η ενημέρωση και η προληπτική γνώση. Ξέρουμε ότι σε κάποιους άλλους τομείς υπάρχουν άλλες νομοθεσίες και ότι γίνεται αξιολόγηση της νομοθεσίας Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο αυτή η αξιολόγηση και μετά να δούμε κατά πόσον ε, χρειάζεται αλλαγή της νομοθεσίας αυτής. Για το τι είναι η διαβούλευση, για παράδειγμα, από ό,τι άκουσα υπάρχουν διάφοροι ορισμοί. Και σίγουρα λοιπόν υπάρχει περιθώριο βελτίωση στο σημείο αυτό. Στην παρούσα λοιπόν φάση να δούμε κατά πόσον υπάρχουν αρκετά εργαλεία για να γίνουν αναδιαρθρώσεις, κατά πόσον είναι χρήσιμο να κινηθούμε προς την κατεύθυνση νομοθετικής πρότασης. Δεν τολμώ στην παρούσα φάση να αποφανθώ να γίνει πρώτα μια αξιολόγηση και μετά με την σωστή ενημέρωση να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις. Thank you. Uh, I'll give the floor to... Ευχαριστώ. Τερίας Κομοντίνη Κατσία από το ΕΛΚ, Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, φαίνεται ότι όλοι συμφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ύψη προτεραιότητα στην πρόθεση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Πώς θα συμβάλλετε εσείς ε, ώστε τα εκπαιδευτικά συστήματα να συμβάλλουν στη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Πώς θα συμβάλλετε στην κινητικότητα των νέων, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, αλλά και στην απασχολησιμότητά τους. Σε ό,τι αφορά την εγγύηση για τους νέους ε, που σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει ακριβώς την ανεργία των νέων, σημειώνουμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014 μόνο δύο κράτη-μέλη άρχισαν να χρησιμοποιούν τα σχετικά κονδύλια. Το πρόβλημα δεν είναι η διαθεσιμότητα κονδύλιων, αλλά ο αργός και αναποτελεσματικός τρόπος εκταμίευσης του από τα, του από τα κράτη-μέλη. Πώς ε, σκοπεύετε να λύσετε αυτό το πρόβλημα? Σας ευχαριστώ η εκπαίδευση και η αγορά εργασίας και η καλύτερη αντιστοιχία που θα πρέπει να υπάρχει είναι ένα πρόβλημα αυτό και θα πρέπει να μας απασχολήσει όντω Αποτελεί άλλωστε και πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό, της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να γίνει αυτό πιο έντονα από ό,τι στο παρελθόν. Και νομίζω ότι αυτό δεν έχει μόνο συμβολική σημασία, αλλά η αρμοδιότητα για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση Δεν είναι συμβολικό ότι όλες αυτές οι αρμοδιότητες που άπτονται των θεμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης έχουν μεταφερθεί στην Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν θα πρέπει να διστάζουμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με τόλμη. Ξέρουμε ότι ενδεχομένως να, υπάρχουν, να υπάρχει κάποια αντίσταση από τους εκπαιδευτικούς αλλά ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση των ενηλίκων θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει καλύτερη αντιστοιχεία. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν καλύτερη ενημέρωση και έτσι να προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τις εγγύησεις για την νεολαία. Συγγνώμη, την πρωτοβουλία για την ε, απασχόληση των ε, νέων. Δώσαμε την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να υποβάλουν γρήγορα λειτουργικά προγράμματα η Ιταλία, η Γαλλία, η Λιθουανία, η Ισπανία έχει υποβάλει σχετική πρόταση. Και φυσικά χρειάζεται χρόνος για να αξιολογηθούν τα προγράμματα αυτά, αλλά να μην ξεχνάμε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει την εργασία τα κράτη-μέλη. Και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπάρχουν διάφορα προγράμματα από την προηγούμενη περίοδο, το Youth Action Program θα πρέπει όλα αυτά να εναρμονιστούν και να φροντίσουμε ο νέος προϋπολογισμός, τα νέα μέσα να αξιοποιηθούν με αποτελεσματικό τρόπο για τους σωστούς σκοπούς για να γίνουν οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά μια παροχή διάστασης νέας για τους νέους. Ευχαριστώ. Το λόγο τον έχει η Μαρία Ζωά Ροντρίγκες για σοσιαλιστές. Αυτή ακρόαση τελειώνει. Κύριε Τάισεν, χρειαζόμαστε δεσμεύσεις σαφείς από εσά. Εδώ είμαι. Σαφείς δεσμεύσεις από την πλευρά σας. Είμαστε όλοι σίγουροι ότι η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κρυθεί από τη δυνατότητα που θα έχει πραγματικά να μειώσει την ανεργία και την ανεργία των νέων, πραγματικά να μειώσει την ένδια και την ένδια των παιδιών και να ελέγξει πραγματικά το κοινωνικό ντάμπινγκ. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να πολεμήσετε για μια οικονομική πολιτική υποστήριξης. Να πολεμήσετε για ισχυρότερους κοινωνικούς στόχους στη στρατηγική Ευρώπη του 2020, στις συστάσεις κατά χώρα, στη βιομηχανική πολιτική και στις επενδυτικές δέσμες μέτρων και χρειάζονται πιο μεγάλη κοινωνική α, στόχη όσον αφορά την Ευρωζώνη, στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ερώτηση. Από τους αντιπροέδρους σας, τους συναδέλφους, Καϊτάνεν και Ντομπρόφσκι, ποιες, ποιους όρους θα ζητήσετε να επικρατήσουν, ποιες συνθήκες να επικρατήσουν για να τα πετύχετε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Είμαι πεπισμένη ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξουν αποτελέσματα. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν ε, μετρήσιμοι στόχοι στο βαθμό του δυνατού. Για να δούμε κατά πόσο έχει αποτελέσματα η πολιτική μας. Η δομή της ε, Επιτροπής, όπως την όρισε ο Ζαν Κλοντ Juncker, είναι μια δομή όπου θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των, κρατών, των ε, Επιτρόπων. Δεν θα είναι καθένας υπεύθυνο μόνο για την αρμοδιότητά του, άλλο για την βιομηχανία, άλλο για την απασχόληση, άλλο για την ψηφιακή αγορά. Όχι, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Και σε ό,τι αφορά την δημιουργία θέσεων απασχόληση, πρόκειται για ένα καθήκον το οποίο είναι κοινό για όλα τα μέλη του νέου σώματο των επιτρόπων. Πώ θα γίνει αυτό συγκεκριμένα, νομίζω ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ποιο είναι ο προγραμματισμό, όταν θα καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα επενδύσεων θα πρέπει πρώτον καθήκον να είναι να παρευρεθώ και να συνδράμω με όλα τα μέσα που έχω στη διάθεσή μου προκειμένου να υπάρξει απασχόληση των νέων, να υπάρχουν νέες επιχειρήσεις, να υπάρχουν κοινωνικές, κοινωνική επιχειρηματικότητα, να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα σε ό,τι αφορά το εξάμεινο, την Ευρωπαϊκή Νομισματική Οικονομική Ένωση, θα συνεργαστώ με τον συνάδελφο για να υπάρξει σωστός συντονισμός και προκειμένου να φροντίσουμε να χρησιμοποιηθούν επαρκείς κοινωνικοί δείκτες και να έχουν ειδικό βάρος, γιατί ως τώρα θεωρούνταν κάτι μάλλον συμπληρωματικό, βοηθητικό αυτοί οι κοινωνικοί δείκτες. Τους κοιτούσαμε αλλά δεν τους χρησιμοποιούσαμε. Νομίζω ότι είναι βασικό, όπως και οι οικονομικοί δείκτες. Εφόσον υπάρχουν οικονομικοί δείκτες, θα πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών και να συμπεριληφθούν αυτά στις ανά αναχώρα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πιο σημαντικό καθήκον μου, αλλά θα υπάρξει καλά συνεργασία. Υπάρχει αυτή η διάθεση για συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και σας διαβεβαιώ ότι αυτό θα κάνω και εγώ. Thank you. Ευχαριστώ. Σαβίνε Βερχέιεν για το ΕΛΚ στην Επιτροπή Πολιτισμού. Υποψήφια επίτροπε, τα κράτη-μέλη που έχουν εισαγάγει το διπλό σύστημα επαγγελματική κατάρτιση συνήθω έχουν χαμηλά επίπεδα ανεργίας των νέων. Παρόλο που ίσω να μην ταιριάζει να αντιγράψουμε το σύστημα για όλα τα κράτη-μέλη λόγω των πολύ διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων όπω προαναφέρατε, αυτό δείχνει ότι μια έγκαιρη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση θα βοηθήσει να ξεπεραστεί η ανεργία των νέων. Τι μέτρα θα λάβετε για να ενισχύσετε τη σχέση μεταξύ εκπαιδείας και επιχειρήσεων. Στα καθήκοντά σας θα προωθήσετε το διπλό αυτό σύστημα σαν βέλτιστη πρακτική στην Ένωση. Και το δεύτερο τμήμα της ερωτήσεως αφορά την εκπαίδευση των ενηλίκων. Ποια σχέδια έχετε όσον αφορά την επίσημη εκπαίδευση παραμόντως στο μικρό, στο πρόγραμμα Ρούμβικ με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό και πώς θα προωθήσετε και τις ίπιες δεξιότητες και την εκπαίδευση των ενηλίκων που ε, στηρίζονται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφε. Η τι εκπαίδευση, είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε το ζήτημα αυτό, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο, μία μέθοδος την οποία γνωρίζουμε όλοι ότι έχει ιδιαίτερα στατικά αποτελέσματα. Έχει αντίκτυπο, λειτουργεί και οδηγεί τον κόσμο στην αγορά εργασίας, δίνει μια καλή εκπαίδευση, αλλά και μια αυξημένη ευκαιρία για προσχώρηση στην αγορά εργασίας. Ξέρετε ότι, και το είπατε και εσείς άλλωστε, ότι οι καταστάσεις διαφέρουν. Δεν υπάρχει μία ενιαία λύση για όλους, αλλά εδώ μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον και γι' αυτό νομίζω ότι στο πρόγραμμα Erasmus Plus είναι πάρα πολύ σημαντική η πτυχή της διαβίου μάθησης και της εκπαίδευσης των ενηλίκων. Μέσω διάθεσης λοιπόν των μέσων αυτών, των ταμείων αυτών, οι εμπλεκόμενοι φορείς σε επίπεδο κράτους μέλους μπορούν να εξηγούν οι μεν στους δε πώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που έχουν, πώς διαμορφώνουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, πού είναι τα δυνατά και τα δύναμα σημεία τους. Και μαθαίνοντας λοιπόν ο ένας από τον άλλον, μπορούν τα κράτη-μέλη να πετύχουν ό,τι χρειάζεται για τις απαραίτητες καινοτομίες. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να, χρησιμοποιούμε, να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις ευκαιρίες αυτές. Είναι χρήματα τα οποία πιάνουν τόπο. Είμαι λοιπόν υπέρμαχος του συστήματος αυτού εκμάθησης και εκπαίδευσης και ξέρω ότι εδώ και χρόνια έχει αποτελέσματα αυτό το σύστημα της εκπαίδευσης και θα πρέπει και χώρες που δεν χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό να δουν πώς μπορούν να το εντάξουν στις δομές τους για το θέμα της εκπαίδευσης των ενηλίκων. Εδώ θεωρώ ότι έχουμε υπερβολικά λίγες πρωτοβουλίες. Υπάρχουν ε, προϋπολογισμοί και κονδύλια τα οποία δεν αξιοποιούνται. Υπάρχει benchmark 15% και είναι 10% μόνο ε, το ποσοστό του κόσμου που τα χρησιμοποιεί τα προγράμματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να παρατρύνουμε τα κρατημέλη να ενισχύσουν τα θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, να τα καταστήσουν πιο αποτελεσματικά και πιο προσβάσιμα. No Thank you. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η Βερόνικα Λόπε Φοντανιά, που είναι και η τελευταία μας ομιλήτρια από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Τίσεν, είμαι η τελευταία ομιλήτρια από την ομάδα μου και θα ήθελα να εκφράσω και δημοσίως την ιδιαίτερη χαρά μου για την ακρόαση που είχαμε, γιατί είστε εξοικειωμένοι με τα θέματα και είναι γνωστός ο αγώνας σας για την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και υπέρ των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Ελπίζω να συνεργαστούμε στενά για να ξαναμπούμε στο δρόμο της υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής του 2020 προκειμένου να καταλήξουμε σε μια πιο δίκαιη κοινωνία που θα έχει και κάποια αηφορία. Χαίρομαι ιδιαιτέρως για την πρότασή σας να αποκτήσει πιο κοινωνικό χαρακτήρα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτό διεκδικεί και η Επιτροπή μας. Επίσης, ως προς το στόχο της μείωσης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, θα ήθελα να σας υποβάλω δύο ερωτήσεις, παρόλο που σχεδόν τα έχετε καλύψει όλα. Τι μέτρα θα προτείνετε για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και δεύτερον, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Πρόσβασης ή Προσπελασιμότητας για τους αναπήρους. Ακόμη εκρεμεί το θέμα αυτό. Θα το προωθήσετε και μάλιστα με σχετική ταχύτητα. Ευχαριστώ. Eh, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Η κοινωνική διάσταση του Ευρωπαϊκού εξαμήνου. Δεν μπορούμε παρά να το τονίσουμε αυτό επανελειμμένως, γιατί έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Μπορείτε να υπολογίζετε και σε μένα και σε όλους τους άλλους επιτρόπους. Έχουμε κατανοήσει το καθήκον μας αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσον υπάρχουν οι σωστοί κοινωνικοί δείκτε. Υπάρχουν κοινωνικοί δείκτε οι οποίοι χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά. Θα πρέπει να λάβουν πιο πολύ ειδικό βάρο. Θα πρέπει να του αξιοποιήσουμε καλύτερα. Δεν λαμβάνουμε μόνο γνώση των κοινωνικών δείκτων. Θα πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένε δράσει στα πλαίσια των συστάσεων αναχώρα. Μπορεί να διαμορφωθεί με πιο κοινωνικό τρόπο το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πώ μέσω Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Από τη στιγμή που γίνονται οι μελέτες μέχρι τις συστάσεις αναχώρα, σε όλη τη διαδικασία πρέπει να υπάρχει συμμετοχή και εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων και των εθνικών κοινοβουλίων. Γιατί αυτά θα πρέπει να φροντίσουν να πηγαίνουν καλά τα πράγματα και σε επίπεδο κρατών μελών, σε ό,τι αφορά τους προϋπολογισμούς, για παράδειγμα. και σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσουμε να μάθουμε πιο πολύ εμένα από τους δε. Για τους αναπήρους, ζητάτε συγκεκριμένη νομοθεσία. Ξέρω ότι έχει τεθεί συγκεκριμένο αίτημα από ένα εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος, ε, αναπήρους, ένα εκατομμύριο σαν, σαν πρωτοβουλία πολιτών πριν καν δημιουργηθεί αυτή η πρωτοβουλία. Το Κοινοβούλιο έλαβε σοβαρά την πρωτοβουλία αυτή την απέστειλε στους προέδρους των ομάδων. Ξέρω ότι υπάρχει σχετική προετοιμασία και προπαρασκευαστική εργασία. Πολύ ευχαρίστω θα ενημερωθώ και θα το θέσω ως προτεραιότητά μου μόλις ολοκληρωθεί η νομοθετική πρόταση να, να φτάσει στο Κοινοβούλιο και να κοιτάξουμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά θέματα προσπλασιμότητας από αναπήρους. Να δημιουργηθεί ένας, μια νέα αγορά για υπηρεσίες και προϊόντα προκειμένου να είναι πιο φθηνά και πιο καινοτομικά. Γιατί ξέρουμε όταν υπάρχει εσωτερική αγορά υπάρχει και πιο πολύ ανταγωνιστικότητα και αυτό αποτελεί καλό κίνητρο για μεγαλύτερη καινοτομία το οποίο και με τη σειρά του θα ωφελήσει τους αναπήρους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής και των άλλων Επιτροπών που έκαναν προετοιμασία και που υπέβαλαν ερωτήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, κάλυψαν ευρύ φάσμα και τις απίθυναν στην κυρία Τάισαν. Θα ήθελα να καλέσω την υποψήφια επίτροπο να προβεί σε μια σύντομη δήλωση, 4 με 5 λεπτά, και να αναφερθεί στα στοιχεία εκείνα που δεν σας επέτραπη να αναφέρετε όταν είχατε να απαντήσετε σε πολύ περίπλοκες ε, ερωτήσεις σε δύο λεπτά. Κυρία Τάισον. Ελεύθερα διατυπώστε κάτι τόσο ώστε να ολοκληρωθεί αυτός ο γύρος ερωταπαντήσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε και αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, επίσης, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για όλες τις ερωτήσεις σας και για την ενδιαφέρουσα ανταλλαγή ιδεών που είχαμε σήμερα και σας διαβεβαιώ για ένα πράγμα. Αν τελικά με υποστηρίξετε και αν μου δείξετε εμπιστοσύνη, θα μετατρέψω τα λόγια μου σε δράση, σε πράξεις Κατά τη διάρκεια της προσπάθησα να σας δείξω ποια θα είναι αυτή η δράση που θα αναλάβω μαζί με σας, με τα κράτη-μέλη και με τους κοινωνικούς εταίρους. Η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επενδύσει σε οικονομική ανάκαμψη και στην προώθηση της απασχόλησης. Θέλουμε να επιστρέψουν εκεί που θέλουν δουλειά σε θέσεις εργασίας, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, να βελτιώσουμε την κινητικότητά τους. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την μέγιστη δυνατή κοινωνική προστασία και για τους εργαζόμενους ανθρώπους και τους μη εργαζομένους και θέλουμε να αντικοπήσουμε τη μάχη κατά της ένδυας. Στόχος μας, καλές και υγιείς συνθήκες εργασίας, θα καταπολεμήσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ και άλλες καταχρήσεις και θα πολεμήσουμε για δίκαιες και ίσες δυνατότητες στην αγορά εργασίας. Αυτή είναι η σαφής στόχη που έχουμε καθορίσει. Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, θέλω να χρησιμοποιήσω πλήρως τα διαθέσιμα μέσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινητοποιήσει μέχρι 300 δις ευρώ για επενδύσεις και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ο προπολογισμό μου αντιστοιχεί περίπου στο 10% του συνολικού ευρωπαϊκού προπολογισμού. Με αυτά τα χρήματα θα προσπαθήσω να πετύχω τους στόχου που ανέφερα, να δημιουργήσουμε θέσει απασχόλησης, να ενισχύσουμε την κοινωνική προστασία και να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Η εγγύηση για τους νέους θα είναι από τις βασικές μου προτεραιότητες και θέλω αυτό το μέσο να εφαρμοστεί πλήρω από όλα τα κράτη-μέλη χωρίς καθυστερήσεις. Στόχος μας προσμετρήσιμα αποτελέσματα διαρκείας. Η απασχόληση και η κοινωνική πολιτική θα αποτελέσουν σαφέστερο, πιο ξεκάθαρο τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν τι αναγκαίε μεταρρυθμίσει. Θα κριθούν βάσει των κοινωνικών του επιδόσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη φιλοδοξία να κινηθεί ενωμένη σαν ομάδα υπό την ηγεσία του Jean-Claude Juncker. Θα συνεργαστούμε και με το Κοινοβούλιο και βέβαια και με τα κράτη-μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους κατανοούμε ότι αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα και μπορούμε να πετύχουμε μόνο αν τα αντιμετωπίσουμε μαζί. Αν σε πέντε χρόνια μπορούμε να πούμε ότι σήμερα η Ευρώπη έχει περισσότερες απασχόλησεις, έχει λιγότερη φτώχεια, τότε θα ξέρουμε αγαπητοί συνάδελφοι και μόνο τότε θα γνωρίζουμε ότι πραγματικά κάναμε τη διαφορά για το λαό. Και όπως είπα και στην αρχική μου παρουσίαση για το λαό δημιουργούμε την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι για τους λαούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Once again, thank you. Uh, Σας ευχαριστώ κυρία Τάισεν εκ νέου. Ευχαριστώ όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην υποβολή των ερωτήσεων. Η συνεδρίαση των συντονιστών θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών για να αξιολογήσουμε την ακρόαση από τις 1 μέχρι τις 2 στην ASP 5G2. Η συνεδρίαση των συντονιστών για την αξιολόγηση των ερωτήσεων και απαντήσεων 1 με 2 στην ASP 5G2. Σας ευχαριστώ όλους. Γεια σας.